Okay, dear colleagues, good morning. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλή σας μέρα. Για το σημείο 5 της ανακοινώσης του Προέδρου δεν έχω ανακοινώσεις. Θα ήθελα όμως ε, να απευθύνω ένα καλωσόρισμα τον κύριο Κλίντ, τον πρώην συνάδελφο. Καλώς μας ξαναήρθατε. Όπως ξέρετε, έχει ξαναέρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή αυτή που για χρόνια ήταν μέλος και στο παρελθόν. Χαιρόμαστε που ξαναβλέπουμε. Έχουμε τις ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις για την κοινωνική έκθεση, αλλά αργότερα. Έχουμε ένα εκρεμές θέμα για την οδηγία για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έχουμε κάποιες καλές ειδήσεις, αλλά όχι ακόμη αργότερα. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 7 και θα ήθελα να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιο επίτροπο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Αγορών. Καλώς ήρθατε κύριε Ντομπρόφσκη. Έχουμε τον τρίτο και τελευταίο ε, διαρθρωμένο διάλογο με τον Αντιπρόεδρο για το 2017 και άσχετα με τις αρμοδιότητές τους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και όλα τα υπόλοιπα που σας ανέφερα. Ε, σήμερα θέλουμε να επικεντρωθούμε και σε αυτό το σημείο βέβαια, αλλά, αλλά φυσικά τα μέλη είναι ελεύθερα να διαμορφώνουν τις ερωτήσεις και το περιεχόμενό τους. Όπως ξέρετε, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια φιλόδοξη ανακοίνωση για την Τραπεζική Ένωση και θα υποβάλει και το πακέτο για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Έχει ξεκινήσει και μια διαβούλευση για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ε, θα συνταχθεί και έκθεση σχετικά και ε, ένα άλλο πακέτο μέτρων Οπότε βρισκόμαστε σε μια σημαντική στιγμή από νομοθετική άποψη. Προσπαθούμε να διεκπαιρεώσουμε, να οριστικοποιήσουμε σημαντικές νομοθετικές προτάσεις και να ε, αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Όταν βέβαια γνωρίζουμε ότι πρόσφατα υποβάλαμε μια σειρά ε, πολύ σημαντικές προτάσεις για το CCP, τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους, το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιδοτικό Προϊόν ε, και ούτω καθεξής, οπότε ε, οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι πλούσιοι από νομοθετικής απόψεως ε, και τις χρηματοπιστωτικές εταιρείε και ούτω καθεξής, αλλά δεν θα πω τίποτα άλλο προς το παρόν. Πολύ χρήσιμο λοιπόν που περνάμε σε αυτή την ε, κρίσιμη φάση των εργασιών μας με το διαρθρωμένο διάλογο με τον Αντιπρόεδρο τον Πρόσκη στον οποίο και δίνω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, καταρχήν να σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση να συζητήσουμε τις εργασίες μας, να συζητήσουμε τις εργασίες έτσι να είναι πιο ανθεκτικός ο χρηματοοικονομικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είδαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης, ένα σωστά λειτουργών ε, χρηματοοικονομικός τομέα είναι κεφαλαιόδης για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση αλλά και την ανάπτυξη. Είχαμε ένα δομημένο διάλογο για το θέμα αυτό τον Ιούνιο. Η οικονομική κατάσταση τη Ελλάδας έχει βελτιωθεί, της Ευρώπης έχει βελτιωθεί έκτοτε. 2,6% θα είναι ο ρυθμό ανάπτυξη για φέτο και στο 1,2% θα είναι πλέον το μέσο έλλειμμα ενώ ε, η ανεργία ε, είναι στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 9 ετών. Είναι ε, αυτή η τάση ενθαρρυντική, όμως η οικονομία μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις. τα επίπεδα δημοσίου και ιδιωτικού χρέου εξακολουθούν να είναι υψηλά και δεν υπάρχουν επαρκεί ε, μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες μέσω βιώσιμης και ε, συμπεριληπτικής ανάπτυξης και βεβαίω έχουμε ακόμα κενά στο χρηματοοικονομικό μα σύστημα. Όπω είπε ο πρόεδρο Γιούνκερ, θα πρέπει να ενισχύσουμε το ενιαίο νόμισμα για να μπορεί αντιμετωπίσει ε, απρόλεπτες προκλήσεις. Έχουμε την Κεφαλαϊκή Ένωση, την Τραπεζική Ένωση. Αυτές ε, είναι διαδικασίε που μπορεί να μα βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο αυτό. Θα μα βοηθήσει επίση να μπορούμε να απορροφήσουμε πιο εύκολα τα σοκ της κρίσης, να προστατεύσουμε καλύτερα τους φορολογούμενους ε, από το να πληρώνουν για τα λάθη του τραπεζικού τομέα και θα μειώσει το κίνδυνο ε, αναταραχών στην Οικονομική Νοσηματική Ένωση. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα που μας παρέχει αυτή τη στιγμή για να ολοκληρώσουμε αυτό που έχουμε ταχθεί να κάνουμε. Αυτό το Κοινοβούλιο έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα να συζητήσουμε λοιπόν μαζί τρεις ε, στόχους κλειδιά από τώρα έως το τέλος της εντολής. Πρώτα απ' όλα να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση και το πλαίσιο του τραπεζικού τομέα γενικότερα. Δεύτερον, ε, η οικοδόμηση της, νέα της νέας ε, κεφαλαϊκής αγοράς και επίσης το θέμα της βιώσιμης, του βιώσιμου χρηματοοικονομικού τομέα. Θα ξεκινήσω από το τραπεζικό. Έχουμε ήδη κάνει πολύ δρόμο λείπει ο τρίτος πυλώνας του τραπεζικού τομέα, το σύστημα ε, ασφάλειας αποταμιεύσεων ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσπαθούμε να φτάσουμε σε συμφωνία για αυτό το σημείο κλειδί. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, ε, αυτό απορρέει από την αρχική μας πρόταση το 2015. Αυτή εξακολουθεί να ισχύει η πρόταση. Ε, Βεβαίω έχουμε διαπιστώσει ότι τα τελευταία δύο έτη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος αλλά όχι αρκετά γρήγορα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δοθεί μια νέα όθηση για να φτάσουμε σε συμβασμό και να ολοκληρωθεί η συμφωνία κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία. Παράλληλα, θα πρέπει να μειώσουμε περαιτέρω του κινδύνου στον τραπεζικό τομέα. Το πακέτο του Νοεμβρίου 2016 περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα για να συμπεριληφθούν εθνικά πρότυπα ε, για τη μείωση των κινδύνων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θέλω να συγχαρώ τους δύο εισηγητές για την πρόσφατη πολιτική συμφωνία σε ό,τι αφορά ε, τον τραπεζικό τομέα, το πρότυπο 9 ε, για τις αναφορές ε, και το θέμα της έκθεσης. Τα υπόλοιπα στοιχεία του πακέτου θα ολοκληρωθούν σύντομα, έτσι ώστε να φτάσουμε σε πολιτική συμφωνία των τομότερο δυνατόν. Επίσης θα πρέπει να επιταχύνουμε την τάση μείωσης των ε, κόκκινων δανείων μη εξυπηρετούμενων την ερχόμενη άνοιξη θα υποβάλουμε ένα πακέτο μέτρων επ' αυτής της βάσης. Μεταξύ άλλων θα περιλάβει και ένα blueprint ε, για τις εθνικές ε, εταιρείες διαχείρισης ε, περιουσιακών στοιχείων αλλά και το θέμα των δανείων που μετατρέπονται σε εξυπηρετούμενο. εξυπηρετούμενα. Αυτό αποτελεί μέρος της πρότασης για την αδιάστρωση και της δεύτερης ευκαιρίας για τους επιχειρηματίες που, που σας παρουσίασε ο συναδελφός μου να μπορέσουμε να φτάσουμε γρήγορα συμφωνία. Προσπαθούμε να βρούμε επίση λύσει έτσι ώστε να λύσουμε το θέμα των sovereign bonds. Εδώ παρακολουθούμε τι προσπάθειε που γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα κρατικά ομόλογα. Αυτά τα μέτρα όλα μαζί είναι ένα φιλόδοξο πακέτο για να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση αυτές οι εργασίες αποτελούν μέρος ε, μιας γενικότερης προτεραιότητα, προτεραιότητας ώστε να ενισχυθεί η Οικονομική Νομισματική Ένωση σε στενή συνεργασία με τους συνάδελφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτές τις δύο προτάσεις τις οποίες θα υποβάλουμε στις 6 Δεκεμβρίου. Μια της πρωτοβουλίες αυτές έχει να κάνει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας θα μπορούσε να μεταφερθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει μια νέα λειτουργία ε, στα πλαίσια και του Ταμείου Ενιαίας Εκαθάρισης. Πέρα από τον τραπεζικό τομέα όμως πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και σε ό,τι αφορά τα παράγωγα, την αγορά παραγόγων. Τα CCPs ε, ε, παρουσιάζουν συστημικό κίνδυνο για το χρηματοοικονομικό τομέα, έχουν και όλο και πιο καταλαμβάνω όλο και περισσότερο χώρο. Υπάρχουν τρει προτάσει ε, για το θέμα αυτό για να ενισχύσουμε την οικονομική σταθερότητα Ταυτόχρονα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, να αποφύγουμε οποιαδήποτε νέο κατακαιρματισμό. Θα συνεχιστεί η συνεργασία με τους εισηγητές για αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, να πει ο κύριος Φον Βάιτσεκερ, ο κύριος Βαν Λάντεν και η Χούμπνερ για την παρακολούθηση των CCP τελευταία. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει υποστήριξη από το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και τώρα θα περάσω στην κεφαλαία αγορά και την κεφαλαϊκή ένωση. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τις πρόσφορε συνθήκες για καλύτερη χρηματοδότηση πραγματικής οικονομίας και μεγαλύτερη ροή χρημάτων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια προηγμένη ένωση αγορών περισσότερο από ποτέ. Μάλιστα, ήδη προωθούμε το, το σχέδιο δράση του 2015 και μάλιστα τον επόμενο μήνα υιοθετήσαμε την πρόταση για διαφανείς διαδικασίες εξακρίβωσης ταυτότητας και επίσης έχουν απλουστευτεί και τα σχετικά ενημερωτικά έντυπα και από κοινού θα έχουμε μία πιο φιλόδοξη Ένωση Κεφάλαιο Αγορών. Θέλουμε καλύτερη ε, πρόσβαση και επιλογή των πελατών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Μάλιστα έχουμε προτείνει τον Ιούνιο ένα ευρωπαϊκό σήμα για, την, για το νέο πανευρωπαϊκό προϊόν ατομικής συνταξιοδότησης που είναι ένα απλό προσιτό προϊόν που πληρεί τις διαδικασίες και τα δικαιώματα του καταναλωτή, αφορά τους ε, χαμηλότοπου λογαριασμού και θα είναι ένα προαιρετικό προϊόν που θα συμπληρώνει τα υπόλοιπα. Και μάλιστα Ευχαριστώ που η κυρία Σοφίνφελτ ε, έδωσε προτεραιότητα στο θέμα αυτό της εκθεσή της. Επίσης, ε, στα συνοριακές πληρωμές και στις ε, διατραπεζικές συνήθειες με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προτείνουμε του χρόνο νέους κανόνες ώστε να πληρώνονται χαμηλότερε προμήθειε από του Ευρωπαίου όταν μεταφέρουν χρήματα εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή παίρνουν χρήματα από αυτόματα μηχανήματα. Και ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που στηρίζει το σχέδιο δράση για τις χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε προ τον καταναλωτή. Επίση, επεξεργαζόμαστε μια πρόταση για τι αρχέ του επόμενου έτου, για να άρουμε τα εμπόδια από την ε, διασυνοριακή μεταφορά κόδηλιών χωρίς μάλιστα να μειώσουμε τη προστασία για τους επενδυτές και με έμφαση στην εποπτεία. Θα αλλάξουμε μάλιστα τη χρηματοδότηση των, των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για να προωθείται καλύτερα η εποπτική σύγκληση και να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις. Κάτι που θα βοηθήσει την σωστή παρακολούθηση και εφαρμογή των αποφάσεων, ισοδύναμων αποφάσεων, με σεβασμό την αρχή της επικουρικότητας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εποπτεία αφορά συγκεκριμένου στοχευμένου κλάδου και στι αρχέ του επόμενου έτου θα υποβάλουμε και ένα νέο πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα. Ε, Αξιοποιώντα κάποια θετικά στοιχεία εθνικών ρυθμίσεων. Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα των προσπαθειών και εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθούμε, προσπαθώντας μέχρι το 2019 να διαμορφώσουμε τις σωστές ε, προϋποθέσεις και όρους αγοράς με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, προκλήσεις ε, όπως η βιώσιμη χρηματοδότηση και η σταθερότητα χρηματοπιστωτική θα πρέπει ήδη να από, από σήμερα να προετοιμαστούμε τη, στην αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. Γιατί σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική τεχνολογία, θέλουμε να γίνουμε σημαντικό παγκόσμιο παράγοντα. Οπότε πρέπει να έχουμε παρόμοιο, ένα σύστημα παρκού παρακολούθηση και μάλιστα για τι αρχέ του επόμενου έτου θα υποβάλουμε σχετικό σχέδιο δράση. Θέλουμε πανευρωπαϊκή νομοθεσία για τέτοια χρηματοδότηση και δανεισμό και επίσης ε, Θέλουμε να προωθήσουμε τις ε, πληρωμές μέσα στο διαδικτύο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα και για την οδηγία, την αθερμένη οδηγία για τι άδειε. Ε, θα έχουμε στενή διαβούλευση με του ενδιαφερόμενου για να ενισχύσουμε την ασφάλεια των ε, γραμμικών πληρωμών, των πληρωμών στο διαδίκτυο και να έχουμε ειδικά συστήματα εξακρίβωση ταυτότητα πάνω από κάποιο κατόφλι, όπω ισχύει σε κάποιε χώρε, και να εξασφαλίσουμε ασφαλέ περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών ε, υπηρεσιών πληρωμών, όπω ε, προσφέρονται από τι τράπεζε χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Οι νέε προδιαγραφέ θα εξασφαλίσει σωστέ προποθέσει και ε, υπό τον όρο τη ρητή στην κατάθεση του πελάτη. Ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και μια μετάβαση προ μια οικονομία με χαμηλέ εκπομπέ άνθρακα. Αυτό δίνει ευκαιρία και στο χρηματοπιστωτικό μα κλάδο, αρκεί να έχουμε τι σωστέ προποθέσει και συνθήκε για να γίνουμε μαγνήτη φιλοπεριβαλλοντικών επενδύσεων με την κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση σχετικών προγραμμάτων. Και αυτό θα αποτελέσει ε, κεντρικό θέμα τη επόμενη Συνόδου Κορυφή για τη χρηματοδότηση του κλίματο στο Παρίσι και περιμένουμε την έκθεση τη ομάδα υψηλού επίπεδου για, για τι αρχέ του επόμενου έτου. Και με βάση τι στάσει αυτέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει ένα σχέδιο δράση για τη βιώσιμη και φιλοπεριβαλλοντική χρηματοδότηση στις αρχές του επόμενου έτους. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, ε, θέλουμε μια πλήρη ένωση κεφαλαγορών, ε, γιατί έτσι θα διαμορφώσουμε ένα ανθεκτικό ε, χρηματοπιστωτικό σύστημα που χρειάζονται οι πολίτε και οι επιχειρήσει και προσβλέπω στη δική σα συνεργασία για να υλοποιήσουμε την αναμενόμενη πρόοδο και να διεκπαιρεώσουμε αυτό το σημαντικό έργο κατά τη διάρκεια της δικής μας θητείας. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Πλούσιο το μενού, πολλά τα ελέη, τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. το psd δύο παραδείγματι που θα μας απασχολήσει και για την ε, εποπτεία, για το διάλογο. Αλλά για να δούμε τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι. Κυρία Σαντέχ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για τα λόγια σας για μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Αγορών, μια πιο ενοποιημένη Ευρωπαϊκή ε, Χρηματαγορά. Θα μας απασχολήσει αυτό ο επόμενος μήνας ασφαλώς και έχω τα ερωτήματα για τις επενδυτικές επιχειρήσεις καταρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να σκοπεύει να κάνει μεταρρύθμιση του εποπτικού προληπτικού ε, συστήματος των ε, επιχειρήσεων αυτών, εκ των οποίων όμως πολλές ε, έχουν έδρα στον Εμένο Βασίλειο. Μήπως με την ευκαιρία αυτής της νομοθετικής πρότασης θα ήταν καλό να αναθεωρηθεί και η νομοθεσία για τις ισοδυναμίες αναγνώριση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που επιτρέπει σε αλλοδαπές επιχειρήσεις να προσφέρουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ ασαφής αυτή η νομοθεσία και στατική πρέπει να πω και δεν επιτρέπει την αντιμετώπιση ε, ρυθμιστικών αποκλήσεων, προστασία ουσιαστική του πελάτη. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Για το crowdfunding Η συμμετοχική χρηματοδότηση λοιπόν θα καλυφθεί από μια νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τις διατάξεις που προβλέπονται και στον κανονισμό ΜΥΦΙΡ βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει αυτή η προστασία. Θέλω να ρωτήσω τι σκοπεύει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πράξει προκειμένου να εξασφαλίσει περισσότερη εναρμόνιση και δυνατότητα για διασυνοριακή παροχή αυτών των υπηρεσιών της ε, συμμετοχικής χρηματοδότησης. Κύριε Στομπρόφκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρώτη ερώτηση. αναθεώρηση της προληπτικής αντιμετώπισης των ε, επιχειρήσεων. Είναι υπό προετοιμασία σχετική νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή οι κανόνες για την προληπτική εποπτεία αυτών των επιχειρήσεων που αφορούν ιδίως όμως τράπεζες είναι στο σχετικό κανονισμό ελέγχου ε, των επενδυτικών κεφαλαίων και τη σχετική οδικία. και άρα τις επενδυτικές επιχειρήσεις δεν τις ε, καλύπτει. Απλώς τώρα προτείνουμε ένα καθεστώς το οποίο ε, θα καλύπτει όλες τις επενδυτικές επιχειρήσεις που έχουν συστημική σημασία με βάση το επιχειρησιακό τους μοντέλο και στοχεύουμε στην επαρκή κάλυψη των κινδύνων, την προστασία του ανταγωνισμού και το σεβασμό των ε, αρχών της, κοινής, ε, της νομισματικής ένωσης. Σημαντικές λοιπόν επενδυτικές επιχειρήσεις, συστημικά συστημικές και λόγω του αντικειμένου τους και λόγω του μεγέθους τους θα πρέπει να παραμείνουν σε αυτό το σύστημα ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει υποπτία και για τις μεγαλύτερες τράπεζες από τον SSM και την, μέσα από την Τραπεζική Ένωση. Το ερώτημα τώρα για την ε, αναγνώριση, την ισοδυναμία στο ΜΕΦΙΤ. Είμαστε όντως σε μια φάση προετοιμασίας. και ετοιμάζουμε ένα έγγραφο που θα παρουσιάζει τις θέσεις μας για τις ισοτιμίες μετά το Brexit. Ένα σημαντικό θέμα που αφορά επίσης τις ισοτιμίες έχει προβλεφθεί να υιοθετηθεί ένα σύστημα ισοτιμιών ενώπιον των πιο σημαντικών ε, αρχών, ε, μάλλον ισοτιμιών επιχειρήσεων των κύριων δικαιοδοσιών. Και αυτό βέβαια αφορά κυρίως ε, Ηνωμένες Πολιτείες και Ελβετία στον αρχικό σχεδιασμό και ταυτόχρονα θέλουμε και να διευκρινίσουμε την αντιμετώπιση των ε, μετοχών που δεν ανήκουν στη ζώνη του ε, ΕΟΧ. Επομένω, θα υπάρξει αυτή η προσαρμογή και πρέπει να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία για τη συμμετοχική χρηματοδότηση, crowdfunding. Θα παρουσιάσει στη Μεσοπρόθεσμη Αναθεώρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ε, ναι, μία πρόταση για τη συμμετοχική χρηματοδότηση και με τη FinTech και με τις ενώσεις χρηματοπιστωτικών αγορών. Προβλέπετε αυτό. Θα γίνουν οι σχετικές διαβουλεύσεις, κυρίως με στόχο την προστασία των, της αξιοπιστίας των πλατφορμών συμμετοχικής χρηματοδότησης, ώστε αυτή η χρηματοδότηση του crowdfunding να μπορεί να περνά και τα εθνικά σύνορα, δηλαδή να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό αυτό της ε, ενιαίας αγοράς και ιδιαίτερη έμφαση θα δώσουμε στην ανάπτυξη ενός συστήματος αδειοδότησης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα απαιτεί από κάθε κράτος μέλος διαφορετική χορήγηση άδεια, έτσι ώστε αυτές οι πλατφόρμες να μπορούν να αναπτύσσονται και πέραν των συνόρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Μεταξύ των νομοθετικών φακέλων που έχουμε εξετάσει στα πλαίσια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης των Κεφαλαιογορών υπάρχει και το κείμενο για το νομισματικό ταμείο που θα ρεθεί ισχύ στην αρχή του επόμενου έτους με βάση τις δημιουργίες που αναλάβουμε στο G20 και το Συμβούλιο χρηματοοικονομικής σταθερότητας ε, για να αποφύγουμε τις κινδύνους ε, του ραν. Ξέρετε ότι προσπαθήσαμε να μειώσουμε τα, τις ΙΝΑΒ, τα ταμεία αυτά τα οποία έχουν ε, έτσι έλλειψη ρευστότητας που έχουν αυτή την τάση ξαφνικής απόσυρσης τους υποχρεώσαμε είτε να γίνουν ε, συνάβ δημοσίου χρέους είτε να γίνουν ε, ταμεία χαμηλής πτητικότητας. Από ό,τι φαίνεται όμως υπάρχει μια πρακτική στην αγορά όλο και πιο διαδεδομένη σε κάποια κρατημέλη που, λέγεται, ε, που ονομάζεται share cancelling. Επιτρέπει λοιπόν σε αυτά τα ταμεία να στα σταθερά τις ε, καθαρές αξίες όταν έχουν αρνητική απόδοση και έτσι ε, να μην μετατρέπονται ε, σε ε, οχήματα μικρής πτυτικότητας. Αυτό το παράθυρο ε, μήπως θα αποτελέσει νέα πηγή αστάθειας μαζί με την ΕΣΜΑ σκοπεύεται να απαγορεύσει αυτή την πρακτική που ουσιαστικά παρακάμπτει και το πνεύμα και το γράμμα του κειμένου του νομοθέτη και επιτρέπει ε, στα πλαίσια του μοντέλου αυτού αυτό που θελήσαμε να καταργήσουμε με βάση το προηγούμενο μοντέλο. Και αυτό είναι κατά και του, της διαφάνειας και της ρευστότητα. Τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε έτσι ώστε να είναι πιο αξιόπιστο το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέναντι ε, στις ε, ακρότητες του shadow banking ε, που είναι η πρώτη μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, ευχαριστώ για το ερώτημα για τα money market funds βέβαια γνωρίζουμε το θέμα αυτό είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε αυτό το συγκεκριμένο θέμα στο οποίο αναφερθήκατε εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι η πολιτική συμφωνία στην οποία έχουμε φτάσει ε, διαφυλάσσεται αυτό σημαίνει ότι αυτά τα ταμεία υπόκειται σε κρατικούς κανόνες και δεν μπορεί κάποιος να παρακάμψει τους κανόνες αυτούς. Όμως όπως είπα σίγουρα θα εξετάσουμε πιο λεπτομερώς ε, το ζήτημα αυτό και θα επανέλθουμε. Okay. We'll do it quickly. Ναι, τι άλλα μέτρα, ε, τι άλλες προτάσεις ε, σκοπεύετε να πάρετε για την αντιμετώπιση του shadow banking. αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ναι, ακούστε για το shadow banking. Αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τον κίνδυνο ε, που παρουσιάζουν αυτές οι νέες πρακτικές και είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Thank you. Case Ευχαριστώ, Κυρία Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε που ήρθατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το επιτελείο σας και κυρίως ε, το, την ομάδα σας ε, για την ε, εταιρεία για τη οδηγία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων που πραγματικά ε, η ομάδα σας προσπαθεί να διορθώσει κάποιες ε, αδυναμίες που επισημάναμε μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής και πραγματικά είναι αξιέπαινη γι' αυτό. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες ε, αδυναμίες που εντοπίζουμε στα θέματα CME. Έχουμε δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες και μάλιστα στην τελευταία τριμερή διάλογο για τα προσπέκτους και για την τιτλοποίηση διαπιστώσαμε τι προσπάθεια έγινε για τις λεπτομέρειες και μας ενοχλεί ότι εντοπίζουμε κάποιες ασυνέπειες που ήδη εμφανίζονται και μάλιστα πριν την θέση σε εφαρμογή αυτών των νομοθετικών προτάσεων. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις και η ταξινόμηση της τιτλοποίησης εντοτήτων ε, ειδικού σκοπού SSP ως κεντρικών αντισυμβαλωμένων δεν ε, συνάδει με τις πρόσφατες συμφωνίες μας στον κανονισμό STS. Επίσης μια άλλη ασυνέπεια είναι ε, στην οδηγία για τα προσπέκτους κάναμε τεράστια προσπάθεια για να δούμε ποιος είναι ο ρόλος των προσπέκτους αυτών ώστε κάποιες ε, ε, αρμοδιότητες να περάσουν από τα STA στον ΕΣΜΑ. Και στην αναθεώρηση ήδη έρχεται αντιφατικές προτάσεις αυτά με αυτά που έχουμε αποφασίσει ό,τι αφορά την ανάγκη σταθερότητας και αυστηρών καρών που απαιτεί η αγορά στο δρόμο προς την εφαρμογή. Είναι πολύ σημαντικό ε, να ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις ήδη σε θέματα που έχουν διεκπαιρεωθεί. Γιατί τέτοιου είδους ε, υπονομεύουν το σχέδιο CME. Ε, αναγνωρίζεται το πρόβλημα και κρίνεται σκόπιμη την αντιμετώπιση του. Φυσικά θα πρέπει να εξασφαλιστεί, εξασφαλιστεί συνέπεια και συνοχή μεταξύ των διαφόρων ε, τμήματων του χρηματοπιστωτικού οικοδομήματος και των σχετικών κανονισμών και αν εξετάσουμε ιδιαίτερα τις οντότητες ειδικού σκοπού, όπως προτείνει η οδηγία ΕΜΙΡ και η μάλιστα η αναθεώρηση της, του κανονισμού ΕΜΙΡ σε ό,τι αφορά τη τυπλοποίηση των STS, τηρούνται οι αποφάσεις που ελήφθησαν στα πλαίσια του κανονισμού για την Οπότε η συμφωνία που έγινε για την ταξινόμηση ε, στην οδηγία για την, ταξι... την παραμένει και τα θέματα της ισοτιμίας ε, και ε, οι κίνδυνοι συναλλάγματος δεν περιλαμβάνονται. Επίσης, το lateral margining λαμβάνονται υπόψη και κάποιες επικουρικές εγγύσεις. Σε ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικές και, τους χρηματοπιστωτικούς και μη χρηματοπιστωτικούς αντισυμβαλόμενους, αυτό συζητήθηκε εν μέρη στο Συμβούλιο και είμαστε ανοιχτοί και προς τη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Και, άλλη καινούρια συνάδελφος. Κυρία Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον κύριο Ντομπρόφσκης που είναι εδώ σήμερα. Όπως και ο προκάτοχός μου εδώ στην έδρα αυτή την κοινοβουλευτική ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τη FinTech, τον, το χρηματοπιστωτικό τομέα που χαρακτηρίζεται από νέες ε, εξελίξεις από την ε, από το υπολογιστικό νέφος, ε, από την τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί τον άνθρωπο να τον βάλουν ε, σε δεύτερη μοίρα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν μια βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τους ε, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και με τρόπο ώστε να μην είμαστε εκτεθειμένοι σε αδυναμίες του κυβερνοσυστήματος. Γιατί όσο περισσότερο στηριζόμαστε στον έφος ε, και τους αλγορίθμους, τόσο περισσότερο είμαστε εκτεθειμένοι σε χρηματοπιστωτικούς κινδύνους. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. Το αναφέρατε κι εσείς, είναι ένα θέμα που απασχολεί και το προσωπικό σας. η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι ένα από τα καθήκοντα ε, στα οποία έχουμε δεσμευτεί εμείς ως Επιτροπή. Πώς λοιπόν εσείς αντιμετωπίζετε τους κινδύνους της ε, κυβερνοασφάλειας στις διάφορες προτάσεις σας για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Και επίσης η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να κάνει μια συλλογική προσέγγιση στην αντιμετώπιση του χρηματοπιστωτικού κινδύνου, περιορίζοντας τους κινδύνους για τις αγορές και τον καταναλωτή ταυτόχρονα. Ευχαριστώ. Thank you. Υπάρχει βέβαια η ε, ομάδα κρούσος, η Task Force για τη FinTech της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξετάζει ακριβώς αυτές τις εξελίξεις τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες νέες δυνατότητες αλλά και κίνδυνοι που μπορεί να ε, αναφαίνονται. Η κυβερνοασφάλεια ασφαλώς είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολεί ιδιαίτερως. Στην κυβερνοασφάλεια πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν περιορίζεται μόνο στη FinTech, γιατί ε, έχει να κάνει και με τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Είναι ένας κίνδυνος για τους πάντες. Γιατί οι υπάροχοι των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στηρίζονται πολύ στην, ε, στον κυβερνοχώρο για την ενημέρωσή τους προκειμένου να προσφέρουν τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και άρα πρέπει να έχουν ε, ασφάλεια από τους κινδύνους της πληροφορικής. Αυτό είναι γνωστό σε όλους και υπάρχουν και οι εδρεωμένες πρακτικές ασφάλειας. Για τη fintech συγκεκριμένα όμως, μια από τις κύριες αρχές που ακολουθούμε είναι η τεχνολογική ουδετερότητα, δηλαδή ανεξαρτήτως της τεχνολογίας που επιλέγεται για την παροχή της υπηρεσίας, εμείς μεριμνούμαστε να προσφέρεται επαρκές επίπεδο ε, προληπτικών διασφαλιστικών δικλείδων και προστασίας του καταναλωτή ή πελάτη. Αυτό είναι απαραίτητο λοιπόν. Να περιλαμβάνει και την ασφάλεια. Ευχαριστώ κύριε Παπαδημούλης. Good Καλημέρα κύριε Ντομπρόσκης. Θα μιλήσω ελληνικά. Πρώτη φορά κύριε Αντιπρόεδρε στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πριν από όλα για τη χώρα μου την Ελλάδα. Πριν από ε, λίγες ημέρες η Κομισιόν έδωσε στη δημοσιότητα τις εκτιμήσεις της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Εκεί προβλέπεται ε, οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα για τα έτη 2018 και 2019 της τάξης του 2,5% και περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, η Ελλάδα υπεραποδίδει στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς αποδίδουν και τα μη παραμετρικά μέτρα που αφορούν περιορισμό κρατικής πατάλης, περιορισμό φοροδιαφυγής, με αποτέλεσμα και να υπερβαίνει τους συμφωνημένους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά και να δίδει η κυβέρνηση ένα σημαντικό κοινωνικό μέρισμα ενισχύοντας τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν ακραία κατάσταση φτώχειας. Και στην Ελλάδα, ξέρετε, είναι έντονο αυτό το φαινόμενο. Επειδή σε λίγες μέρες κατεβαίνουν τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ντομπρόφσκης, με βάση την εκτίμηση που έχετε και τις πληροφορίες που έχετε, θεωρείτε εφικτό το στόχο που ακούω ότι έχει τεθεί να έχουμε staff level agreement στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου και ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης στο Eurogroup της 22ης Ιανουαρίου του 2018 η έγκαιρη ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης από ό,τι ξέρω είναι και για την ελληνική κυβέρνηση και για την Κομισιόν ένας σημαντικός στόχος προκειμένου να έχουμε οριστική έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 2018. Θα ήθελα την εκτίμησή σας σε αυτά. Uh, okay. Uh, on uh, Greece. Ναι, λοιπόν, για την Ελλάδα. Ακούστε, βεβαίως, η ελληνική οικονομία ανακάμπτει. Αυτό το επιβεβαίωσε και το επιβεβαίωσαν οι οικονομικές προβλέψεις του φθινοπόρου. Αναμένεται όντως ε, υψηλός δημός ανάπτυξης, μείωση της ανεργίας. Ε, σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό τομέα, επίσης διαπιστώνουμε ότι αποδίδει και υπεραποδίδει η προσπάθεια της Ελλάδας ό,τι αφορά τους στόχους τους δημοσιονομικούς και ο στόχος του 1,75% πλεονάσματος ε, ε, έχει επιτευθεί και επειδή ακριβώς υπήρξε υπέρβαση του στόχου ένα σκέλος ε, αυτού των περαιτέρω χρημάτων θα διατεθούν, θα διατεθούν ως κοινωνικό μέρισμα αυτή η προσέγγιση ευθυγραμμίζεται με το μνημόνιο και η Ελλάδα επίσης είναι πολύ κοντά σαν να πετύχει και τους στόχους για το δημοσιονομικό πλεόνασμα του χρόνου. Αναφερθήκατε στη βελτίωση της ίσπραξης φόρων ε, και αυτό είναι ένας τομέας όπου συνεργαζόμαστε στενά με τις ελληνικές αρχές. Ε, ενισχύουμε και τις φορολογικές αρχές τις ελληνικές με την, ε, με την όποια απαραίτητη τεχνική συνδρομή και συμφωνούμε με την αξιολόγηση ότι γρήγορη ε, ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης θα είναι ένα θετικό μήνυμα ότι δηλαδή το πρόγραμμα προχωράει κανονικά και αυτό μπορεί να ε, βοηθήσει την Ελλάδα να προετοιμαστεί για μια ε, επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Δεν θέλω τώρα να δεσμευτώ σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, υπάρχουν μια σειρά προαπαιτούμενα ε, που πρέπει να πληρώνται Πάντως ε, στο τέλος του του έτους, στην αρχή του επόμενου, είναι απολύτως εφικτό ε, να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση. Αυτό το χρονοδιάγραμμα έχουμε και εμείς κατά νου. Ευχαριστώ. Μάλιστα, πολύ ωραία. καλέ ειδήσει. Ο κύριος Ορτασούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Η ομάδα μου ανησυχεί ακόμη τα μάλα με τα προβλήματα το too big to fail και μετά από τις πενταετής προσπάθειες ε, τις νομοθετικές, ελάχιστα έχουν βελτιώσει τα, τα κεφαλαία τους και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα οι τράπεζες. Και μάλιστα για το benchmark στο οποίο ε, επιμείνατε, ε, τέτοια μοντέλα είναι ε, πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και δεν δίνουν μια αξιόπιστη εκτίμηση κινδύνων. Και μάλιστα η τροποποίηση των κανόνων των τελευταίων μηνών και οι σχετικές προτάσεις προσέκτουσαν σε αντιδράσεις ε, των κυβερνήσεων και το τραπεζικό κόστος ε, είναι πολύ ψηλότερο από την απόδοση γιατί οι επενδύσεις θεωρούνται ε, ρηψοκίνδυνες. Και έτσι υπάρχει λιγότερη διαφοροποίηση και λιγότερη εμπέδωση στον τραπεζικό τομέα και λιγότερη σταθεροποίηση σε σχέση με το παρελθόν. Και μάλιστα Έχουμε υπερβολικό αριθμό τραπεζών και οι εκθέσει δείχνουν ότι χρειάζεται κατεπηγόντω μεταρρύθμιση. Δεν θα πρέπει να, γίνουν κάποιες, ε, να είχαν γίνει ήδη κάποιε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια, παρά τις προσπάθειες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκρούει σε ένα τείχο ε, πολιτικής απροθυμίας. Πότε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχοληθεί με αυτόν τον ελέφαντα στο δωμάτιο, κάτι που όλοι γνωρίζουν αλλά αποφεύγουν το, το πρόβλημα των μεγάλων τραπεζών που είναι υπερβολικά μεγάλες για να πτωχεύσουν. Δεν πρέπει να επιλύσετε επιτέλου το πρόβλημα για να μην χρησιμοποιούνται κονδύλια των φορολογουμένων για τη διάσωση τραπεζών και του τραπεζικού συστήματος. Ο κύριος Δομπρόφσκης. Ω προ την πρώτη σα ερώτηση για το too big to fail. Όπως ξέρετε, υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος. Ένας τρόπος είναι μια διαρθρωτική ε, μεταρρύθμιση των τραπεζών. Μια τέτοια προσπάθεια, όπως ξέρετε, κόλλησε ε, για χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πρώτη ευρωπαϊκή Επιτροπής είχε θετηθεί ήδη από το 2014. Το Συμβούλιο συμφώνησε στη Γενική Προσέγγιση το 2015. Αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ε, προώθησε αυτό το θέμα και τελικά αποσύρθηκε η σχετική πρόταση. Βέβαια το πρόβλημα παραμένει, αλλά στο μεταξύ προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Με άλλους τρόπους όμως. Για παράδειγμα, με την ενίσχυση των προληπτικών απαιτήσεων και είχαμε σχετικούς κανονισμούς και προωθήσαμε ένα πακέτο για μέτρα μείωσης του κινδύνου πέρυσι τον Νοέμβριο. Αναφερθήκατε σε κάποια εσωτερικά μοντέλα γι' αυτό. Προτείναμε υποχρεωτικό συντελεστή μόχλευσης ως μηχανισμό προστασίας για τα εσωτερικά μοντέλα των τραπεζών. Και μάλιστα και στην Επιτροπή της Βασιλείας ε, αυτό το θέμα που συζητείται είναι το Output Floor. Εκεί συζητούμε το πώς επηρεάζει την ευαισθησία στους κινδύνους. Υπάρχουν ακόμη μερικές απορίες και ερωτηματικά. Πάντως θα συνεχιστεί η δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση. Και υπάρχουν και άλλα ε, θέματα που βοηθούν τη σταθερότητα. Το τελεστής χρηματοδότηση, για παράδειγμα, για να αποφευθούν οι αναντιστοιχίες μεταξύ πιστώσεων και δανεισμού ή επενδύσεων. Και μία από τις προτάσεις μας πέρυσι στο πακέτο μεταρρυθμίσεις των τραπεζών είναι το ΤΛΑΚ δηλαδή η συνολική ικανότητα απορρόφησης κινδύνων για τις ε, συστημικά σημαντικές παγκοσμίω τράπεζες. Ε, καλύπτουμε και την περίπτωση αυτή σε περίπτωση που χρειαστεί εξηγίαση. Και μάλιστα εμείς ξεπερνούμε τις παγκόσμιες προδιαγραφές γιατί έχουμε ελάχιστες απαιτήσει για τα MRL, τα, τις επιλέξιμες υποχρεώσεις και τα διαθέσιμα κεφάλαια. Υπάρχουν πολλά στοιχεία λοιπόν που συνάδουν στη μείωση των κινδύνων και στην αντιμετώπιση του προβλήματος του too big to fail με άλλους τρόπους. Και αυτό και απευθύνουμε έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιταχύνει τις συμφωνίες ε, για το πακέτο μέτρων για τη μείωση των κινδύνων που έχει επιτάπητος και εξετάζει. Όντως ε, Είχαμε χάσει την ευκαιρία στο παρελθόν και μάλιστα τη συνέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το 3% μόχλευση είναι το ισοδύναμο περίπου της προηγούμενης πρότασης. Ελπίζω να μην περάσουμε από το too big to fail στο too small to survive. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και αυτό αναζητούμε. Μια ισορροπημένη λύση στο πακέτο μέτρων για τη μείωση του κινδύνου. Ο Μάρκο Βάλλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και περιμένω να βάλω το ακουστικά σα. Θα επανέλθω με την ερώτηση του κυρίου Ορτασούν για την απάντηση της Επιτροπής. Δεν είναι επαρκής, δηλαδή δεν νομίζω ότι θεωρείται σκόπιμο από πλευρά σας να επανέλθει με μία πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν αρκετές επικρίσεις σχέση με την Τραπεζική Ένωση στο βαθμό που έχει εξαντληθεί αυτή σε ένα bail-in και δεν προστατεύει τον καταναλωτή, κάτι το οποίο έχουμε δει και στην Ιταλία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες όπου καλείται ο πελάτη τράπεζα, ο να συμβάλλει στη διάσωσή της. Δεν μπορεί να υπάρχει λοιπόν χωρί αυτή την απαραίτητη διάκριση επαρκή τραπεζική ένωση. Οι μεγάλες τράπεζες ξέρουμε ότι αντιτίθενται όμως στην ε, περαιτέρω πρόοδο της, χρημα... της ε, Τραπεζικής Ένωσης και γι' αυτό θα πρέπει να δείξει πυγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι να προχωρήσει. Επίσης, θέλω να ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι μία διαχείριση πιο υπεύθυνη θα ήταν σκοπιμότερη προκειμένου να μην χάνονται τόσα χρήματα με την ε, κερδοσκοπία η οποία εν τέλει οδηγεί τις τράπεζες δυσκολίες και μετά βέβαια στον Μπέιλιν και μετά στην ανάγκη να συμβάλλει ο πολίτης, ο καταθέτης, τις ε, απώλειες για να καλυφθούν οι απώλειες μιας ε, ανεύθυνης διαχείρισης. Δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε ή θα μπορούσε να γίνει ακόμη μία αξιολόγηση ως προς το γεγονός ότι ορισμένες τράπεζες έχουν ε, χαρτοφυλάκια, διακρατούν χαρτοφυλάκια διαφορετικών επιπέδων και ποιότητας και ότι άρα θα μπορούσαν να ε, καταστούν σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνες οι καταστάσεις αυτές και άρα θα έπρεπε να υπάρχει ένας τρόπος ε, να διαφυλαχθούν ε, τουλάχιστον να διαφυλαχθεί η ρευστότητά τους. Ευχαριστώ. Ντομπρόφσκης. Ακούστηκαν αρκετές ερωτήσεις. Αλλά επαναρχόμαστε με το too big to fail. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο επίπεδο αυτό. Από το 2014 με την πρόταση της Επιτροπής που είχα εγώ υπευθύνη μου για αρκετά χρόνια, νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει με άλλες πρωτοβουλίες για να ε, αντιμετωπίσουμε το ίδιο θέμα με διαφορετικά μέσα. Τα οποία περιέγραψα στην απάντηση που έδωσα στον κύριο Ουρτασούν. για, τις, ε, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καταρχάς και την ε, διαβούλευση που έγινε στον ε, ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Έχουν όντως ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις που θα κρατήσουν μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου, ίσως 6 Δεκεμβρίου και μετά γίνεται η συζήτηση στον SSM, στο μηχανισμό, με βάση τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης. Και των πληροφοριών που θα αντιληφθούν από αυτήν. Σε σχέση με τις δράσεις της Επιτροπής, εμείς ακολουθούμε μία εντολή που ορίζει ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η δράση μας αναπτύσσεται σε διάφορες κατευθύνσεις, τις οποίες περιέγραψα. Έχουμε παραδείγματι ένα σχέδιο για τις εθνικές εταιρείε διαχείρισης ε, ε, ενεργητικού, το πλαίσιο, τις πρωτοβουλίες για την ε, δευτερογενή αγορά, για τις δευτερογενείς αγορές ε, των μη εξυπηρετουμένων δανείων, για προληπτική δράση, με, διάφορες, με διάφορα στάδια, η παραδείγματι στοχευμένη διαβούλευση για νομοθετικά, νομοθετικές παρεμβάσεις προληπτικά. Ταυτόχρονα έχουμε, όπως είπα, μια εντολή μέσα στην οποία εργαζόμαστε. Και οτιδήποτε καταλήξω, οτιδήποτε νέα συμπεράσματα καταλήξουμε, αυτά δεν μπορούν παρά να αφορούν τα νέα δάνεια. Όχι τα παλαιά μη εξυπηρετούμενα. Επίσης για τις ε, τράπεζες επίπεδου 3 και το ενεργητικό τους, γι' αυτό το λόγο έχουμε ακριβώς τρία διαφορετικά επίπεδα δράσης, αφενός μεν τον κανονισμό, όπου σκοπεύουμε τον επόμενο χρόνο να καταθέσουμε προτάσεις. Το δεύτερο επίπεδο που είναι οι εποπτικές ε, δράσεις από τον SSM προς τις τράπεζες και εδώ υπάρχει ένα πεδίο δράσης έναντι της κάθε μεμονωμένης τράπεζας, σε συνδυασμό βέβαια με τις δράσεις και του ε, επίπεδου 1. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Κουαλτιέρη. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλά σχεδιασμένο και ισορροπημένο το πακέτο της Επιτροπής. Κύριος Τσάνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία και κύριε Πρόεδρε, θα θυμάστε ότι πριν από μερικού μήνες έγινε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψε μεταξύ μελών της Επιτροπής μας και του ε, Προέδρου Ντράγκη για, τους, ε, για, για το ενδεχόμενο αποχώρησης από το ευρώ μιας ε, χώρας όπου μας είπε ότι τότε θα παρέμενε υποχρέωση για την απόδοση των υπολείπων του, των χρεωστουμένων, δηλαδή του στόχου 2 ή του επίπεδου 2, ενώ για τον στόχο 2, σε περίπτωση εξόδου για τη Γερμανία, μας είπε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλέπεται από τις συνθήκες. Όλοι Ρένος, το 2012 ο προκάτοχός σας, απαντώντας σε μια γραπτή ερώτηση δηλαδή πρόκειται για επίσημη ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλώνει και σας διαβάζω ότι αν κράτος μέλος Ευρωζώνης αποφασίσει να αποχωρήσει δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 50 της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα θέτει και τέρμα στη συμμετοχή του στο ενιαίο νόμισμα και έτσι λοιπόν απευθύνομαι σε εσάς ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι και σαματοφύλακας των συνθηκών για να ρωτήσω εάν ήταν εσφαλμένη η ερμηνεία του Προέδρου Ντράγκη ο οποίος δεν ε, θεώρησε δυνατή την εξέλιξη αυτή ή εάν στην επίσημη εκείνη απάντηση και ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είχε δώσει λάθος, λάθος πληροφορίες. Τεν του λέμε στα λατινικά, δηλαδή ή το ένα ισχύει ή το άλλο και τα δύο μαζί δεν γίνεται. Ο κύριος Γουαλτιέρη, βεβαίως έχουμε ελευθερία του λόγου εδώ. Μπορείτε να κάνετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Βέβαια είχαμε πει ότι ε, μεγάλο τμήμα της ακρόασης της χθεσινής με τον κύριο Ντράγκη θα ήταν αφιερωμένο στο στόχο 2 και εξε, ε, εξέθεσε τις θέσεις του διεξοδικά. Βέβαια εσείς δυστυχώς δεν ήσασταν παρόν, ε, αν δεν απατώμε, αλλά ε, στο διάλογο αυτό με τους συναδέλφους και την παρουσία του κυρίου Ντράγκη. Λάβαμε την ε, αυθεντική ερμηνεία από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το θέμα αυτό. Αυτό για να είμαστε τόσο ακριβείς και συγκεκριμένοι. Από εκεί πέρα βέβαια έχετε το ελεύθερο να αναφερθείτε σε οποιοδήποτε τμήμα συγκεκριμένης διατύπωσης αποκομμένης από μια μεγαλύτερη παράγραφο και να την ερμηνεύσετε όπως θέλετε, αλλά κατά τα άλλα Μα δεν, δεν είναι θέμα στόχου 2, target 2, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την ευθύνη. Δεν είναι τι θα μας πει ο πρόεδρος. Ε, μα είναι απλό το ερώτημα και όλοι ρε, έχει ήδη απαντήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όντως, είναι δύσκολο να σχολιάσω την ερμηνεία του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας ε, εχθές, αφού δεν μπόρεσα να διαβάσω ακριβώς λέξη προς λέξη τι είπε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει γνωστός μηχανισμός αποχώρησης από την Ευρωζώνη και δεν βλέπουμε να φεύγει καμία χώρα. Άρα δεν υφίσταται στην πραγματικότητα ζήτημα και δεν θα πρέπει να μας απασχολεί. So, do you confirm... Eh? Δηλαδή κύριε Αντιπρόεδρε, εσείς ε, επικυρώνετε την επίσημη απάντηση του, ότι, η επίσημη απάντηση του Όλη Ρέν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ψευδής. Ότι αν αποχωρήσει μια χώρα δυνάμει του άρθρου 50 της συνθήκης φεύγει και από το Γυροζώνη. Μα είναι δεδομένο, λέει ο κύριος Γκουαλτιέρη, ότι δεν μπορεί να φύγει κανείς από το ευρώ χωρίς να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν φύγει από την Ευρωπαϊκή, για να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε ότι υπάρχει το άρθρο 50. Είναι χρήσιμο να το γνωρίζει κανείς. Αλλά η ερώτηση είναι διαφορετική. Εσείς λέτε πώς θα φύγει κανείς από το ευρώ. Και όλοι η Ρέν η απάντηση για το πώς θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν φύγει, αν φύγει κανείς από την Ένωση αποχωρώντας πρώτα από το ευρώ είναι άλλη ιστορία. Δηλαδή, λέει ο κύριος Τσάνη, εσείς Επιβεβαιώνεται ότι έσφαλε ο πρόεδρος Δράγκη όταν είπε ότι δεν μπορεί που δεν, κανείς να φύγει από την, την Ευρωζώνη. Γιατί δεν προβλέπεται από τη συνθήκη. Ο κύριος Γουαλτιέρη απαντά. Ναι, δεν προβλέπεται από τη συνθήκη να ξεχωρίσει κανείς το ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι γνωστό τη πάση αυτό άρα δεν υπάρχει λόγος να το συζητούμε. Καλά, Μάλιτιτς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. για τις προσπάθειες που καταβάλλετε σε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας ότι σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της ε, ε, Κεφαλαιακής Ένωσης ε, θέλετε να αντιμετωπίσετε τα βασικά εμπόδια στην ελεύθερη ροή κεφαλαίων. Και αυτό είναι κάτι που συνδέεται με την δεύτερη ευκαιρία, την αναδιάρθρωση και τις αλλαγές σε πάση ε, ε, στον κανονισμό περί Θα ήθελα λοιπόν για αυτές τις αλλαγές στον κανονισμό για την αφαιρεγγιότητα να σας θέσω ένα ερώτημα. Βεβαίως το 2018 θα μας απασχολήσει το θέμα αυτό. Ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες στα κράτη-μέλη, να το εξασφαλίσουμε αυτό. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκοπεύετε να εργαστείτε παράλληλα για τη δημιουργία δυνατοτήτων στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εξασφαλίσετε εκ των προτέρων μια ομαλή εφαρμογή, μια ομαλή υλοποίηση για να μην έχουμε πάλι διαφορετικές πρακτικές αποκλίνουσες από χώρα σε χώρα όπως συμβαίνει σήμερα με τον κανονισμό αφαιρεγγιότητας που ισχύει. Επίσης πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε κάποια επιμέρους λύση σε ό,τι αφορά τις εταιρείε ε, συστημικής σημασίας αυτά για την αφαιρεγγιότητα και τον σχετικό κανονισμό τώρα κάτι που αφορά το σημείο 3 για την ε, βιώσιμη χρηματοδότηση. Εδώ είναι κάπως παράδοξη η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ καλύτερα από ό,τι αυτά της καινοτομίας. Και τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη start-up. Επίσης ε, τα startup, οι startups δημιουργούν, δημιουργήσουν ε, προβλήματα όταν θέλουν να αλλάξουν κλίμακα. Ε, μπορείτε να υποβάλλετε κάποια πρόταση για το πώς θα ε, ε, δοθούν κίνητρα ε, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις για να επενδύσουν ε, στις ε, startup αυτές σε διάφορα στάδια όμως ανάπτυξής τους για να τους επιτρέψουν όχι μόνο να δημιουργηθούν αλλά και να αναπτυχθούν στη συνέχεια. Ναι, θέσατε μια σειρά από ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, για το δίκτυο σχετικά με την αφαιρεγκαιότητα Αυτό αποτελεί μέρος των εργασιών μας και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το σχετικό σχέδιο δράσης. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα benchmark σε ό,τι αφορά την εθνικό, τα εθνικά πλαίσια αφαιρεγγιότητας για να δούμε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε μέσω συγκεκριμένων συστάσεων ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ε, για να τροποποιηθούν ενδεχομένως τα εθνικά πλαίσια. Επίσης υπάρχουν κάποιες προτάσεις μεταξύ των οποίων η πρόταση για την ε, δεύτερη ευκαιρία και την έγκαιρη αναδιάρθρωση που δίνουν τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης τις επιχειρήσεις ε, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τα δραστηριότητά τους ε, χωρίς ε, η, διαδικασία αφαιρεγκαιότητα να οδηγήσει σε πτώχευση εφόσον βεβαίως συνθήκε συνθήκες βιωσιμότητας. Επίσης θέλουμε να υπάρχει μια επιταχυμένη εφαρμογή από, τα, από τις τράπεζες των collateral είναι κάτι που αφορά όμως μόνο εμπορικά δάνεια ενδεχομένως ε, και αυτό θα μπορούσε να βελτιώσει τα ισοζύγια των τραπεζών. Είχαμε μια δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο και θα υποβάλουμε πρόταση στο πρώτο τρίμηνο του ερχόμενου έτους. Τώρα αναφερθήκατε στη βιώσιμη χρηματοδότηση. Η βιώσιμη χρηματοδότηση, όπως είπα, θα ακολουθήσουμε ε, την τελική έκθεση της ε, ομάδας ψηλού επίπεδου των πυρογνωμόνων με ένα νέο σχέδιο δράση στην αρχή του ερχόμενου έτους. Εκεί θα υπάρξουν μια σειρά πρωτοβουλίες ε, για να μπορέσουμε να κατευθύνουμε τη χρηματοδότηση προς βιώσιμους πράσινους στόχους ε, σε ό,τι φορά τη start-up τώρα, τις ιδιωτικές ε, ε, έχουμε ένα νέο πλαίσιο για το κεφάλαιο κινδύνου και την κοινωνική επιχειρηματικότητα εξετάζουμε τι συμβαίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς μπορούμε ε, ακριβώς να χρηματοδοτήσουμε την ε, ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε διάφορα στάδια για να μπορούν όχι μόνο να ξεκινήσουν να δημιουργηθούν επιχειρήσεις αλλά να μπορούν στη συνέχεια να μεγαλώσουν κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Χώνας Φερνάντες. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε και καλώς ήρθατε στην ΕΚΟΝ. Είστε πρόσδεκτος πάντα. Θα σας θέσω μια ερώτηση για την ανακοίνωση που αφορά την Τραπεζική Ένωση και κυρίως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων, το ΕΝΤΙΣ. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πώς η Ευρωπαϊκή επιμένει στην νομοθετική πρόταση που έχει υποβάλει πριν από δύο χρόνια και προ... προτείνει μία νέα ερμηνεία που αλλοιώνει το αρχικό σχέδιο, την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό πραγματικά μα μπερδεύει. Γιατί με την νέα ερμηνεία που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που στην πρώτη φάση ρευστότητα ε, προσθέτει την αρεσιμότητα, κάτι που δεν είχε στην αρχική πρόταση, και μετά κάνει σαφή μνήμα της διατήρησης της τελικής φάσης με ε, αμοιβεοποίηση αυτής της ε, ε, ασφάλειας καταθέσεων, με κοινή ανάληψη κινδύνων αυτή τη ασφάλεια καταθέσεων. Αυτό έχει προβληματίσει και εμένα και την ομάδα μου. Πώ είναι δυνατόν να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση και λίγο μετά μια τελείω διαφορετική νομοθετική πρόταση, αντιφατική. Και σε ποιο βαθμό επιμένει στη δέσμευσή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φτάσει στην τελευταία φάση τη πλήρη ανάληψη κινδύνου ε, που με βάση την δεύτερη πρόταση έχει αλλοιωθεί. Τώρα, δεύτερη ερώτηση ως προς την ανακοίνωσή σα για την Τραπεζική Ένωση ανακοινώσετε μια πρόταση fiscal backstop, ενός μηχανισμού στήριξης που θα μπορούσε να είναι το MEDER και το ESM για την Τραπεζική Ένωση και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας για τις συζητήσεις που γίνονται στο Eurogroup γιατί πέραν των προτάσεων Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Eurogroup έχει ρόλο στον προσδιορισμό αυτού του μηχανισμού στήριξης ε, fiscal backstop μαζί με το ε, ESM. Πώς βλέπετε επίσης ε, την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον, μελλοντικό πρόεδρο, με τον μέλλοντα πρόεδρο του Eurogroup. Ο κύριος Δομπρόφσκης. Τώρα, για το θέμα της ανακοίνωσης της Τραπεζικής ε, Ένωσης. Η ανακοίνωση αυτή είναι ανακοίνωση όπως λέγεται το όνομά της, δεν περιλαμβάνει νομοθετικές προτάσεις. Μόνο η νομοθετική πρόταση που βρίσκεται επιτάπητος, δηλαδή η αρχική πρόταση του 2017, 15 συγγνώμη, είναι νομοθετική. Η ανακοίνωση είναι μια ανακοίνωση. Και τι κάνει η ανακοίνωση? Προσπαθεί να διευκολύνει τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πτερίγων της νομοθετικής αρχής. Γιατί από το 2015, από την κατάθεση της νομοθετικής πρότασης, δεν είδαμε μεγάλη πρόοδο μεταξύ των ε, δύο νομοθετών. Και επίσης ε, αναφέρθηκαν κάποιες ανησυχίες για την πρόταση για το έντις και την πιθανότητα του ηθικού κινδύνου στο θέμα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων. Γι' αυτό και προτείναμε κάποια στοιχεία προς εξέταση στους ε, νομοθέτες, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το πώς θα ε, εφαρμοστεί πιο σταδιακά το ΕΝΤΙΣ, το σύστημα ασφάλειας καταθέσεων και μία αξιολόγηση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων πριν διαπιστωθεί ε, πώς θα ληφθούν υπόψη, λαμβάνοντας ε, υπόψη και το θέμα του ηθικού κινδύνου. Και η μετάβαση στο, στο στάδιο 2 περιλαμβάνει κάποια απορράψη των σημειών, και κρατά και την τελική φιλόδοξη της πρότασης που είναι απόλυτη ανάληψη κινδύνων ε, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλειας Καταθέσεων. Αυτό είναι ο τελικός προορισμός, η τελική φιλοδοξία που είναι η ίδια και της ανακοίνωσης και της αρχικής νομοθετικής πρότασης. Στο ό,τι αφορά το fiscal backstop, επικεντρωνόμαστε τώρα στο μηχανισμό στήριξης του ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Έγιναν ε, κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις, πρόσφατα μάλιστα, για το θέμα αυτό στο Eurogroup. Και μάλιστα υπήρξε ευρεία στήριξη ώστε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας να είναι μηχανισμός στήριξης του, Ευρωπαϊκού Ταμείου, του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίασης. Και υπάρχει συμφωνία επί της αρχής και με το Κοινοβούλιο πριν από μια τετραετία για τη σύσταση ενός τέτοιου μηχανισμού στήριξης. Ήρθε η ώρα τώρα να δράσουμε και να εφαρμόσουμε αυτό το μηχανισμό στήριξης, τον backstop. Σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο του Eurogroup, αυτό θα το σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι υπουργοί ΕΚΟΦΗΝ θα επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρό τους, τον επόμενο πρόεδρο του Eurogroup. Και ήδη έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις και οι διαδικασίες σχετικά με την εκλογή του επόμενου πρόεδρου του Eurogroup. Ο κύριος Στόλογιαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσει. Η μία έχει να κάνει με την διευκόλυνση που ανέφερε ο πρόεδρος Γιουνκέρ ώστε να διευκολύνει τις χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη να ενταχθούν σε αυτήν. Τι λεπτομέρειες έχετε σε σχέση με το μέσο αυτό. Φερρυπή νέος κανονισμός είναι να προταθεί πιστώσεις θα διατεθούν και επίσης υπάρχουν ε, γιατί τη FinTech ήδη, ακούστηκαν κάποιες ερωτήσεις των συναδέλφων. Ο πρόεδρος Δράγκη είπε ότι το πλασματικό χρήμα δεν είναι στο σχεδιασμό της έκτα, αλλά είναι μια πραγματικότητα στη ζωή των Ευρωπαίων. Έχετε υπόψη κάτι να πείτε ή να κάνετε σε σχέση με το εικονικό νόμισμα. Ντομπρόφσκης. Πρώτη ερώτηση. Όντως, στο πλαίσιο της εμβάθυνσης αυτής της ε, Ονέέ προβλέπουμε την ε, υποστήριξη, την προενταξιακή στην ΟΝΕ για τις χώρες που ετοιμάζονται να υιοθετήσουν το ενιαίο νόμισμα, όπως είπε και ο Πρόεδρος Ιουνκέρ, πρόκειται κυρίως για τεχνική υποστήριξη, που μπορεί όμως να λάβει και ε, χρηματοοικονομικό μορφή για το τμήμα της τεχνικής υποστήριξης. Μπορούμε να βοηθήσουμε στη δουλειά της μεταμόρφωσης των ε, διαφόρων υπηρεσιών με τα προγράμματα που έχουμε για διάρθρωση και μεταρρύθμιση. Επίσης πολύ σημαντικό είναι το ότι δίνουμε το μήνυμα μιας πιο θετικής στάσης ε, ενεργητικής και ε, μεγαλύτερης βούλησης για δράση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως ε, μπορεί ένα κράτος να αποστείλει το μήνυμα ότι ναι, μπορεί ένα κράτος να αποφασίσει να ενταχθεί στο ευρώ ή όχι και τα δύο είναι αποδεκτά, αλλά για τα κράτη τα οποία σκοπεύουν να ενταχθούν στο ενιαίο νόμισμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει το μήνυμα ότι θα έχουν την υποστήριξή της, την ένθερμη. Επίσης, για το ψηφιακό ή εικονικό νόμισμα. Ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και άλλες κεντρικές τράπεζες έχουν δώσει τα μηνύματα. Τα εικονικά νομίσματα δεν συνιστούν νομίσματα με την έννοια της ε, κατανόμων παροχής οικονομικής εγγύησης, οικονομικού αντικρίσματος, δεν έχουν το αντίκρισμα το νομικό. Ε, μπορεί να είναι ένα μέλος μέρο, τμήμα συναλλαγής, ένα ε, μέσων συναλλαγών, αλλά όχι, δεν έχουν νόμιμο αντίκρισμα. Ε, ωστόσο, ταυτόχρονα μας απασχολεί το οικονομικό νόμισμα και στο πλαίσιο της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και στη σχετική οδηγία κοιτούμε να διευκολύνουμε τις αρχές τήρησης και επιβολής του νόμου στον δυνατό και απαραίτητο βαθμό, ώστε να διερευνούν και κινδύνους που ενδεχομένως απορρέουν από εικονικά ή πλασματικά νομίσματα και αν δούμε ότι δεν αρκούν αυτές οι διατάξεις είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και σε συγκεκριμένε προτάσεις. Για ορισμένους τομείς άλλωστε έχουμε ήδη οθετήσει κάποιες ε, διατάξεις. Ευχαριστώ κύριος Φωνβάης Τσέκα. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση ε, των τραπεζών. Ο κύριος Γκούναρ Χέκμαρκ ε, ασχολείται με το θέμα αυτό και πέραν των μέτρων που ελήθησαν ε, για να ε, γίνουν πιο ισχυρέ τράπεζε ε, και πιο ανθεκτικέ, ε, θεωρεί ο κύριος Χάκμαρκ ότι δεν χρειάζεται τέτοια άλλη διαρθρωτική μεταρρύθμιση. Εγώ διαφωνώ. Και η συμφωνία που δόθηκε από την έκθεση Λικάν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκολουθεί να ισχύει. Ποιο έχει δίκιο όμω, χρειάζεται επιπλέον διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζών ή όχι. Έχουμε κολλήσει λίγο εκεί. Έχω μία πρόταση λοιπόν. Γιατί δεν ξανασυγκαλείτε την ομάδα Λικάν για να σας βοηθήσει. Κάναν, συγγνώμη, για να μπορέσετε να αποφασίσετε τελικά και ίσως ε, να υποβάλλετε καλύτερη πρόταση για να επιλύσετε τα κρεμή προβλήματα. Ή μήπω έχει δίκιο ο Γκούναρ Χέκμαρ, ο συνάδελφο, ότι δεν χρειάζεται πια μετά τα μέτρα που έχουν τα ε, μεταρρύθμιση διαφορετική των τραπεζών. Ερωτώ λοιπόν, πρόκειται να ξανασυγκαλέσετε την ομάδα Λικάναν για να λάβετε μια πιο ξεκάθαρη γνώμη και να διαμορφώσετε πιο εμπεριστατωμένη άποψη για το ποιο είναι το σωστό και τι μελιανέστε. Αυτή είναι η πρότασή μου για την διαρθρωτική μεταρρύθμιση των τραπεζών. Σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, την οικονομική, χρηματοοικονομική τεχνολογία. Ε, θα ήθελα να συνεχίσω την ερώτηση του κυρίου Στόλογεν. Έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχαμε συντάξει μια έκθεση ε, και ήμουν και εισηγητής και μάλιστα ζητήσαμε να συγκληθεί μια ομάδα εργασίας ε, ειδική ώστε να προλάβουμε ε, τη σώρευση κινδύνων. Ε, γιατί σκεφτείτε τους κινδύνους στην αγορά bitcoin. Έχει φτάσει, έχει ε, διωκωθεί. Έχει γίνει μια φούσκα αυτή η αγορά του bitcoin. Και πολύ φοβάμαι ότι θα σπάσει κάποια στιγμή αυτή η φούσκα της αγοράς του bitcoin και, και θα επισκιάσει, θα μαυρώσει τη φήμη αυτή της νέας ε, τεχνολογίας. Πότε λοιπόν ε, θα, ομάδα, θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας για τη Strip Technology ώστε να αποφύγουμε ε, τέτοιες καταστάσεις και κινδύνους σαν αυτή της αγοράς bitcoin. Μάλιστα. Για την πρώτη ερώτησή σας, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τραπεζών. Αυτό το ζήτημα απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και πολλά χρόνια. Από το 2014 που υποβάλαμε και την πρότασή μας, θα έλεγα, και μάλιστα και ο προκατοχός μου, ο κ. Χίλ, είχε ασχοληθεί με το ζήτημα. Και εγώ πέρυσι τον Οκτώβριο που ανέλαβα τα νέα μου καθήκοντα, είχα συνάντηση και με την ομάδα διαπραγμάτευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να προσπαθήσουμε να προλιώνουμε το έδαφος και να ξεφύγουμε από αυτό το αδιέξοδο. Προς το παρόν όμως δεν το έχουμε ακόμη καταφέρει. Διαπιστώσαμε ότι δεν σημειώθηκε πρώτος δυστυχώς για το θέμα αυτό της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης των τραπεζών. Έχουμε πέσει σε τείχο. Οπότε, όπως σας είπα και πριν, ε, κάποια από τα στοιχεία για να αντιμετωπιστούν κάποιες ανησυχίες του, της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης προωθούνται μέσω άλλων νομοθετικών προτάσεων. Για το ΤΑΚ, τα ΜΡΕΛ, αυτά είναι επιμέρους στοιχεία του πακέτου της ικανότητας απορρόφησης σημειών ή ε, το ελάχιστε απαιτήσει δύο κεφαλαίων ε, και επιλέξιμων υποχρεώσεων και απασχολούν ε, και την Επιτροπή της Βασιλείας. Τώρα θα σκεφτώ την πρότασή σας για την επανασύσταση της Επιτροπής Λικάναν, της ομάδας Λικάναν και θα μπορούσα να συζητήσω και με τον ίδιο τον κύριο Λικάναν για να μου πει τις απόψεις του για το θέμα αυτό. Τώρα το Digital Distributed Ledger Technology είναι κάτι που το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην ειδική ομάδα εργασίας FinTech της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και μάλιστα έχει ξεκινήσει και ένα πιλωτικό πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για, για την, Ευρω... την διαφανή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χρηματοοικονομικά ζητήματα και μάλιστα στα μέσα Δεκεμβρίου θα ολοκληρωθεί αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και θα έχουμε και μια έμπρακτη απόδειξη για το πώς ε, λειτουργεί αυτό το σύστημα που είναι δημοσίως προσβάσιμο και στο ίντερνετ. Και μάλιστα ε, τα είναι και τα σχετικά έγγραφα, τα τεχνικά και τα επιχειρηματικά. Και από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του πιλωτικού προγράμματος ε, τα είδαμε και τα συζητήσαμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τις αρμόδιους οργανισμούς, την ΕΣΜΑ μεταξύ άλλων και θα συνεχίσουμε αυτό το έργο προσπαθώντας και στον προπολογισμό του 2018 να χρησιμοποιήσουμε ε, ε, να χρηματοδοτήσουμε ένα, ε, πακέτο, ένα, ναι, ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την ηλεκτρονική εξακρίβωση ταυτότητας των εταιριών και φυσικών προσώπων. Έτσι, θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη νέα τεχνολογία και να αποφύγουμε τους κινδύνους που μπορεί να ενέχει. Ο κύριο Νίτερμαϊερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε κύριε Επίτροπε. Ένα γενικό ερώτημα. Συνήθω εξετάζουμε πολύ τεχνικά ζητήματα εδώ, αλλά επειδή πλησιάζει το τέλος της θητεια ε, σιγά σιγά, θα πρέπει να δούμε λίγο και τα αποτελέσματα. Θα ήθελα να αναφερθώ στην στο εμβληματικό πρόγραμμα ε, για φέτος αυτό της Τραπεζικής Ένωσης, της Κεφαλαϊκής Ένωσης, της Συνεργειακής Ένωσης. Ε, θα ήθελα να ξέρω ε, υπάρχει πιθανότητα να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η Τραπεζική Ένωση βεβαίως είναι ένα σημείο κλειδί, είναι και το πιο προβληματικό. Βλέπω την ανακοίνωση ε, της Κομισιόν, ε, είναι σαν να βλέπω ήδη τα εμπόδια μπροστά μου. Τι μπορεί λοιπόν να γίνει για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και πόσες πιθανότητες δίνεται ως το τέλος της θητείας να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, ε, να υπάρξει δηλαδή συμφωνία για την Τραπεζική Ένωση. Τώρα για την Κεφαλαϊκή Ένωση όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να υπάρξει με μεγαλύτερη ισορροπία ε, στον τραπεζικό τομέα, το οικονομικό, όμως αυτό το σχέδιο είναι ακόμα πιο δύσκολο ε, εσείς τι πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να μας παρουσιάσετε σε ένα χρόνο από τώρα. Ποια θα είναι τα απτά, τα ορατά αποτελέσματα. Έχουμε να δώσουμε απαντήσεις, έχουμε να, θα μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε πετύχει κάποιους από τους στόχους που θέσαμε πριν από τρία χρόνια. Ευχαριστώ. Ναι, ακούστε, πρώτα απ' όλα να πω ότι βεβαίως εμείς προφανώς και ελπίζουμε ολοκληρωθούν οι εργασίες, ε, θα ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση και η Κεφαλιακή Ένωση ε, και βεβαίως ε, γι' αυτό εργαζόμαστε και ελπίζουμε να υπάρξει υποστήριξη και από το Κοινοβούλιο προς την κατεύθυνση αυτή. Τα σημεία κλειδιά πάντως για την Τραπεζική Ένωση είναι η μείωση του κινδύνου, το πακέτο για τη μείωση του κινδύνου του περσμένου Νοεμβρίου που υποβάλαμε και έχει ήδη υπάρξει μια πρώτη συμφωνία για τους, ε, τα, τα, τα, όρια έκθεσης, ε, το πρότυπο παριθμών 9 και άλλα. Υπάρχει το ΕΝΤΙΣ ε, και το, το Ταμείο το, το εξυγίανσης και για τις, ε, την κεφαλαϊκή αγορά έχουμε ήδη ολοκληρώσει τα δηλαδή δύο τρίτα του αρχικού σχεδίου δράσης ε, θα πρέπει τώρα να ολοκληρώσουμε την προσπάθειά μας υπάρχουν όμως κοινέ πρωτοβουλίες που έχουν υποβληθεί για ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ε, συνταξιοδότησης θα πρέπει να το δούμε και αυτό επίσης ε, είχαμε μια αναθεώρηση των ε, αρχών των τραπεζικών υπάρχει και μια δράση για, τα, για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λιανικής δίνουμε κυρίως έμφαση εδώ στις χώρες εκτός Ευρωζώνης, ένα πλαίσιο ε, για τα καλυπτόμενα ομόλογα. Υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίες λοιπόν, ευρύτερες. Αναφερθήκαμε στο πλαίσιο αφαιρεγγιότητας ε, και κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία δεν αφορούν την κεφαλαϊκή ένωση ακριβώς, αλλά ε, θα παίξουν ρόλο για την ολοκλήρωση της ένωσης αυτής Οπότε ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστεί μαζί μας έτσι ώστε να σημειώσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη πρόοδο. Ευχαριστώ. Η Περβάνς Μπερέζ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αναφέρατε την πρότασή σας, την πρόταση της Επιτροπής δηλαδή, για την ε, επισκόπηση αναθεώρηση των ευρωπαϊκών ε, αποκεντρωμένων υπηρεσιών. Βρισκόμαστε βέβαια στην ε, εκκίνηση της συζήτησης. Και βλέπουμε ότι, όχι το Συμβούλιο μόνο, αλλά γενικά και οι ίδιοι εμπλεκόμενοι διερωτώνται πώς θα γίνει η διάρθρωση μεταξύ των υφισταμένων δομών ε, διαχείρισης, διοίκησης και των προτάσεων των δικών σας για ένα διοικητικό συμβούλιο. Μπορείτε να διευκρινίσετε καταρχάς τους λόγους για τους οποίους δεν γίνονται αυτές τις προτάσεις. Και δεύτερον, υπενθυμίζω ότι εδώ στο Κοινοβούλιο είχαμε την ευκαιρία σε μια συζήτησή μας να μιλήσουμε με τον Ζάκ Ντελαροζιέρ, ο οποίος είχε ιδιαίτερος επιμείνει στην ανάγκη για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες να υπάρχει διαχωρισμός της εποπτείας και της λειτουργίας. Αυτός είναι ο λόγος των προτάσεων σας. Και αν ναι, τι έχετε να πείτε ως προς τις επικρίσεις ότι περιπλέκει η πρόταση αυτή ιδιαίτερα το θέμα της διαχείρισης, της κυβέρνησης. Ο κύριος Δράγκη, ε, χτες αλλά και άλλοι πριν, έχουν ε, εκφράσει ανησυχίες τους για το δικαίωμα ψήφου που θα μπορούσαν να έχουν σε αυτές τις υπηρεσίες και την εκπροσώπηση. Θεωρείτε ότι είναι ικανοποιητική η κατάσταση. Επίσης, σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις και τις προτάσεις σας ε, για αναθεώρηση, πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν με τις ερωτήσεις τους ε, στο θέμα του bitcoin, του εικονικού νομίσματος. Ε, πιστεύετε ότι οι υπηρεσίες είναι έτοιμες και επαρκώς καλυμμένες, έχουν επαρκή εξοπλισμό στα χέρια τους και μέσα για την αντιμετώπιση αυτών των νέων τεχνολογιών έτσι ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο οργανωμένο με καλή εποπτεία που να αποτρέπει τη χρήση του εικονικού νομίσματος για τη χρηματοδότηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας ή, πες περιπτώσει, να μας εκθέτει σε κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων. Ευχαριστώ, για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Αρχής. Αυτό που προτείνουμε είναι η θέσπιση στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών ε, Διοικητικό Συμβούλιο για να είναι πιο αποτελεσματική η διαδικασία λήψεων αποφάσεων. Και έχουμε κάτι σαν πρόεδρο, δηλαδή και συνέλευση εθνικών εποπτικών αρχών. Γιατί σε σχέση με αυτές τις συνελεύσεις εθνικών εποπτικών αρχών, παρατηρείται μια κάποια τάση προστασίας των εγχώριων συμφερόντων και αποκοπή από τις ε, άλλες δικαιοδοσίες. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι ότι αναθέτουμε σε αυτό το εκτελεστικό συμβούλιο, διοικητικό συμβούλιο, τη λήψη κάποιων συγκεκριμένων αποφάσεων και το διοικητικό το εκτελεστικό σύμβολο λοιπόν έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο αποφάσεων και τις στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνει το ε, Διοικητικό Συμβούλιο, Συμβούλιο Διαχείρισης. Αυτή είναι η πρόταση. Πρόσφατα κατατέθηκε στους συνομοθέτες. Βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε δυνατότητες βελτίωσης ή ενίσχυσης του συστήματος. και βέβαια άλλων συντημάτων που αναφέρεται σχέση με τον ε, SSM κτλ. Α, τώρα για το bitcoin, για το εικονικό νόμισμα, νομίζω ότι αυτό μπορεί να υπαχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο εντολής που προτείνουμε για το fintech, για την εντολή δηλαδή που θα έχει και να καλύπτει και το εικονικό νόμισμα, όπως άλλωστε λέμε ότι μπορεί να καλύπτει και την πράσινη και αηφόρο ή βιώσιμη χρηματοδότηση. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να δώσουμε τα εργαλεία στα χέρια των υποπτικών αρχών που τους είναι απαραίτητα για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και ίσως ένας ευρωπαϊκός κανονισμός να είναι πιο καλά προσαρμοσμένο σε επίπεδο fintech κυρίως, προκειμένου να επιτρέπει μια δράση πέραν των συνόρων. Ε, ευχαριστώ. Ναι, νομοθέτες εμείς είμαστε βέβαια, είναι σημαντικό αυτό. Και με την Επιτροπή θα συζητήσουμε δυνατότητες βελτίωσης. Βεβαίως και υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης, εφόσον το αποφασίσουμε. Αντιλαμβάνομαι πάντως ότι και η Επιτροπή βλέπει πως έχει περιθώριο βελτίωσης. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και βέβαια έχουμε και εξαιρετικούς, εξαιρετικούς ε, εισηγητές. Ο κύριος Χακμαρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον δόκτωρα Φαβάισεγκερ, τον ε, ε, εξέχοντα συνάδελφο που επισήμανε το θέμα το, της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης. Όταν κανείς χάνει τα κλειδιά του, πρέπει να ψάχνει εκεί που θεωρεί ότι το έπεσαν. Ε, πρώτα πρέπει να προσδιορίζουμε το πρόβλημα πριν ε, ασχοληθούμε με τη λύση του, παρά να επινοούμε ή να φανταζόμαστε ότι κάπου υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει ε, η συζήτηση για τους συστημικούς κινδύνους. Είναι κάτι που μας προβληματίζει συνεχώς. Και αν δούμε την παγκόσμια οικονομία, τις ευρωπαϊκές οικονομίες, διαπιστώνουμε ότι ένα από τα προβλήματα είναι ε, η υπερχρέωση. Στην... Στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το ξέσπασμα της κρίσης ε, εντάθηκε το φαινόμενο όχι μόνο της ιδιωτικής χρέωσης αλλά και της χρέωσης του δημοσίου. Και στην Ευρώπη είχαμε παρόμοιο πρόβλημα και λύσαμε το πρόβλημα της υπερχρέωσης ε, αυξάνοντας το δανεισμό. Παρόμοιο πρόβλημα υπερχρέωσης έχουν και κάποιες ασιατικές οικονομίες. Και αυτό ήταν ένα δίδαγμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το συνειδητοποίησαμε την αλληλεπίδραση του χρηματοπιστωτικού με το τραπεζικό σύστημα. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι είναι τεράστιο πρόβλημα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε πολλά κράτη-μέλη. Είναι η έλλειψη των ε, επενδύσεων ε, χρηματοδότησης, γιατί ό, όταν έχουμε χαμηλή ανάπτυξη, τόσο μεγαλύτερος είναι ρυθμός των κόκκινων δανείων. Και έχουμε και άλλους συστημικούς κινδύνους επίσης. Μήπως λοιπόν, βέβαια, μπορείτε να συζητήσετε με τον κύριο Λικάναν και να ρωτήσετε τι γίνεται με τις άλλες εναλλακτικέ προτάσεις που περιείχε η έκθεση και που τις αγνόησε, τις ξέχασε ο διαπρεπής συνάδελφος. Γιατί λοιπόν να μην επεκτείνουμε τη συζήτηση και να συγκεντρώσουμε και νέες απόδειξεις, όχι για τον ίδιο τον κανονισμό, αλλά για να εντοπίσουμε τους συστημικούς κινδύνους να δούμε πού υπάρχουν οι συστημικοί κίνδυνοι και στην παγκόσμια οικονομία και στην ευρωπαϊκή οικονομία και τι πρέπει να κάνουμε για να τους αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι η απάντηση δεν είναι μόνο ε, η επαναφορά στο παλιό πρόβλημα ότι οι τράπεζες παρά είναι μεγάλες. Αυτό είναι πολύ εύκολο και εντάσσεται στην πολιτική ρητορική, αλλά η εμπειρία μας έχει δείξει ότι το πρόβλημα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας δεν ήταν μόνο οι μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες, αλλά οι επενδύσεις στα ακίνητα, οι μικρότερες τράπεζες, οι τράπεζες επενδύσεων και η αλληλεπίδρασή τους και η υπερχρέωση, το βάρος του χρέους. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε μια πιο σύγχρονη συζήτηση που θα στρέφεται προς το μέλλον πιο, πιο ανοιχτή από ότι ε, να έχουμε μια περιορισμένη συζήτηση σε παλιές λύσεις όπως πρότεινε ο συνάδελφος προηγουμένως. Ο κύριος Δομπρόφσκης, δείξατε μια σειρά ζητημάτων. Μερικά αφορούν και μακροοικονομικά θέματα και το χρηματοπιστωτικό κλάδο, ε, το υψηλό επίπεδο χρέωσης και ιδιωτών και του δημοσίου. Αυτό όντως είναι παράγον κινδύνου, το αναγνωρίζουμε και γι' αυτό επικεντρωθήκαμε στη προσπάθεια μείωσης του χρέους και στις ειδικέ συστάσεις αναχώρα αναφερόμαστε ε, στον τρόπο που συσσωρεύτηκαν τα δάνεια και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα με ενυπόθηκα δάνεια, με δάνεια και προσπαθούμε να μειωθεί αυτό το, αυτό το επίπεδο χρέους ε, και αναλύουμε και τους κινδύνους που επιφέρει σε ό,τι αφορά τις τράπεζες ε, και θα μπορούσαμε ίσως να το αντιμετωπίσουμε και με διαφορετικό τρόπο, με κάποια συστήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλούμε για, τον, για το ενιαίο Ταμείο Εξυγίασης, για παράδειγμα. Και επίσης ε, ζητούμε μεγαλύτερη διαφοροποίηση στους ισολογισμούς των τραπεζών. Και αυτό το εξετάζει και το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και εντοπίσαμε ότι η έλλειψη επενδύσεων ε, δημιουργεί πρόβλημα και αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες της πολιτικής μας. Και μάλιστα αύριο που θα υιοθετήσουμε το φθινοπορεινό μας πακέτο της αιτήσεις επισκόπης για την ανάπτυξη θα το αναφέρουμε και εκεί εξετάζονται πολλά σχετικά θέματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων ή το call for evidence που ζητάτε, τη συγκέντρωση τεκμηρίων σε σχέση με τους ε, συστημικούς κινδύνους. Νομίζω ότι έχουμε αντιληφθεί επαρκώς τους συστημικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε. Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να έχουμε πιο διορατικό τρόπο ανάλυσης ε, και στραμμένο προς το μέλλον Δηλαδή να εξετάσουμε και τους υφισταμένους κινδύνους, αλλά να προλάβουμε και κάποιους μελλοντικούς κινδύνους. Για παράδειγμα, ε, νέες εξελίξεις στις οικονομικές, χρηματοοικονομικές τεχνολογίες ή στη συζήτηση για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Οι κλιματικές αλλαγές είναι επίσης πηγή δυνητικά μακροπρόθεσμων συστημικών κινδύνων στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία που θα πρέπει να εξεταστούν και να αναλυθούν. Και μάλιστα με τρόπο διορατικό και στραμμένο προς το μέλλον, όπως είπατε κι εσείς. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ για την υπενθύμηση. μερικά από τα σχόλια και τα δικά μου και ζητήματα που ήθελα να θίξω ήδη απαντήθηκαν και η Περβάνς μίλησε για τις εποπτικές αρχές. Εγώ θα μιλήσω για ένα θέμα που με αφορά μέσα, το θέμα των κεντρικών αντισυμβαλωμένων, των τρίτων χωρών και της εποπτείας. Είναι ένα ζήτημα που παρακολουθώ και σταχθήκαμε υπέρ της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ αντοπίζουμε δύο ή τρία μάλλον θέματα που χρήζουν ε, ανάλυσης. Το πρώτο είναι πώς θα αποφύγουμε την ε, υπερβολικά περίπλοκη διακυβέρνηση. Και έχουμε πολλά θέματα επί τόπου. Έχουμε το, το, το Συμβούλιο των, ε, της ΕΣΜΑ, έχουμε το νέο Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πολλούς φορείς. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα ώστε να απλουστεύσουμε και να εξορθολογήσουμε αυτές τις δομές. Επίσης, διαβάσαμε προσεκτικά τη, γνώμη, τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το άρθρο 22 της τροποποίησης του καταστατικού και αντιλαμβανόμαστε ότι η πρόθεσή σας είναι να δώσετε αρμοδιότητες στην ΕΚΤ αλλά να τις πλαισιώσετε, να τις περιχαρακώσετε για να αποφευχθούν επικαλύψεις με την Ομοθετική αρχή, με την Επιτροπή ή με τις αρμοδιότητες άλλων οργάνων. Φυσικά θέλουμε να διασφαλίσουμε τις νομισματικές αρμοδιότητες της ΕΚΤ και ερωτώ πώς βλέπετε εσείς αυτό το θέμα και ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα πιθανά σφάλματα επικάλυψης ε, που η γνωμάτευσή σας για την τροποποίηση του καταστατικού προσπαθεί να αντιμετωπίσει και να αποτρέψει. Άλλο τραγωνισμός του κύκλου είναι η αναγγελία των ε, κανόνων μηχανισμών ισοδυναμίας με τις τρίτες χώρες, αποφεύγοντας τον κατακαιρματισμό των αγορών. Έχουμε καλές συμφωνίες με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Πιστεύετε ότι κάποιες διατάξεις μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Και τέλος, ε, χαίρομαι και επικροτώ την ε, ισορροπημένη πρότασή σας για τα μη ξυπηρετούμενα δάνεια. Και σε αντίθεση με ό,τι είπε ο συνάδελφος, και το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι διαβουλεύσεις της ήταν σαφέστερες για το τι πρέπει να γίνει από τις ρυθμιστικές αρχές ε, για το πεδίο εφαρμογής. Επίση επίσης, ε, τον προληπτικό μηχανισμό στήριξης και την ανάγκη ε, πιο περιεκτικού πακέτου και δέσμης μέτρων για να ε, καλυφθούν και κάποια θέματα πληρονομικά. Θα ήθελα να ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει ενεργά σε αυτές τις κοινέ προσπάθειες των θεσμικών οργάνων, ώστε και να αντιμετωπιστούν και να μειωθούν αισθητά τα κόκκινα δάνεια και να γίνει κάτι τέτοιο με εύτακτο τρόπο, να αποφεύγοντας ανεπιθύμητες και περιττές συνέπειες. Ναι, ακούστε για το πρώτο ερώτημα για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους ε, και την εποπτεία τρινών χωρών. Η πρόταση υπάρχει, αναγνωρίζουμε δηλαδή ότι αυτά τα CCP είναι όλο και πιο σημαντικά για το σύστημα και παίζουν ρόλο για την οικονομική σταθερότητα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα σύστημα υποπτίας και για αυτούς τους σχετικούς συμβολόμενους ε, τρίτων χωρών εφόσον υπάρχει δυνατότητα αυτών των CCPs να εγκαταστηθούν, να εγκαταστηθούν εντός της ε, ενίας αγοράς. Τώρα για τις δομές ανάπτυξης έχουμε προτείνει μια ισορροπημένη κυβερνητική ε, μάλλον μια ισορροπημένη δομή διακυβέρνησης όπου η Κομισιόν, η ΕΣΜΑ, ε, οι κυβερνήσεις δρούν στα πλαίσια των του τους. Ελπίζουμε ε, αυτή, μια αυτή να είναι μια ισορροπημένη δομή, αυτή προτείνουμε και αυτό φαίνεται και στην πρότασή μας για αναθεώρηση, την αναθεώρηση του άρθρου 22 του καθεστώτος ε, του καταστατικού της Κεντρικής Τράπεζας όπου αναγνωρίζουμε ότι η ΕΚΤ έχει αυτές τις αρμοδιότητες αυτή ήταν και η βάση της απόφασης ε, του δικαστηρίου που απέρριψε τη δυνατότητα της ΕΚΤ να αποφασίσει για ε, τον, ε, την έδρα των τοπικών των κεντρικών αντισυμβαλωμένων. Γι' αυτό λοιπόν τροποποιούμε το καταστατικό με έναν τρόπο όμως που να είναι συνεπής με την πρότασή μας στα πλαίσια του ΕΜΙΡ. να υπάρχει συνέπεια δηλαδή, μεταξύ, μεταξύ των νομοθετημάτων. Τώρα για την διεθνή διάσταση και τις διεθνείς ε, προεκτάσεις. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει έτσι ε, μια κάποια αγωνία από τους διεθνούς εταίρους μας τι επιπτώσεις θα έχει αυτό για τις τρίτες χώρες εμείς είμαστε σαφείς τους ε, διαβεβαιώνουμε ότι αυτό σε καμιά περίπτωση δεν ε, επηρεάζει την ισοδυναμία αποφάσεων. Είμαστε ε, διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με τους διεθνείς εταίρους μας για να αποφύγουμε οποιοδήποτε κατακαιρματισμό της αγοράς. Τώρα, για το NPS, για, για τα μη να δάνεια, τα NPLs, ε, ε, εργαζόμαστε, εργαζόμαστε σκληρά και θα συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο ώστε η προσέγγιση που ακολουθούμε μια προσέγγιση ισορροπημένη που λαμβάνει υπόψη διάφορες πηγές κινδύνου για το οικονομικό σύστημα θα μπορέσει να προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο, τον κ. Ντομπρόφσκης, για αυτήν την εξαιρετικά χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων και τώρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. και ο διάλογος βεβαίως θα είναι συνεχής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα κρίσιμα νομοθετήματα. Ευχαριστώ πολύ.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 με το να Καλημέρα σας και πάλι. Σημείο 8 στην ημερήσια δάταξης. Επισκόπηση κατεξιοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων. Δύο, δηλαδή ένα. Είναι τα θέματά μας με το... και με ένα δεύτερο θέμα στο τελευταίο κομμάτι. Ένα γνωστό RTS. Προδιαγραφές και ασφαλής ενημέρωση, πρόταση της Επιτροπής. Το ιστορικό το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω. Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, συζητήσεις που κάναμε εδώ, ανταλλαγές απόψεων, έντονες εδώ στο Κοινοβούλιο, δέσμευση τη Επιτροπή να τα αναλογιστεί όλα αυτά πολύ προσεκτικά και τώρα μάλλον πλησιάζουμε μια τελική, σε μια τελική πρόταση που θα συνδυάζει διάφορα στοιχεία. Μακάρι, αλλά πρέπει να ακούσουμε με προσοχή. Και τα τελευταία δέκα λεπτά θα μας απασχολήσει το RTS, το άρθρο 7.6 του κανονισμού των ε, τελών συναλλαγών για τις τραπεζικές ε, πιστοτικές κάρτες ζητήματα τα οποία είναι ακόμα σε εξέλιξη και προτιμώ τις ε, δικές μου παρατηρήσεις να τις διατυπώσω μετά αφού ακούσουμε τους ε, συναδέλφους και την Επιτροπή. Έχουμε συμφωνήσει νομίζω ήδη έτσι ότι θα δώσουμε το λόγο πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία και καλωσορίζω. Ραφ και λυπή. από τη ΦΙΝΣ και από την ε, Γενική Διευθυντή Ανταγωνισμού, από την ΕΤΑ, από την ΕΚΤ. Είναι πολλοί οι εκπρόσωποι και δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής πρώτα. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ και είμαι ευγνώμων στην Επιτροπή σας για την ευκαιρία που μας δίνει να συζητήσουμε αυτή τη τεχνική προδιαγραφή για την επιτυχή υλοποίηση του PSD2. Πρόκειται για ένα περίπλοκο νομοθέτημα, δεν το έχετε δει ακόμη. Πολλοί όμως θα γνωρίζουν ότι για το πρότυπο αυτό υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Θέλουμε λοιπόν να αναπτύξουμε το πλήρες δυναμικό της οδηγίας για τις ε, πληρωμές, για τις υπηρεσίες πληρωμών και για την ενοποίηση των λογαριασμών σε αυτές έτσι ώστε να έχουμε στο δυνατόν πιο ασφαλές σύστημα πληρωμών. Όλες οι πλευρές που εμπλέκονται στις συζητήσεις, που ενεπλάκησαν στις συζητήσεις για τη τεχνική προδιαγραφή, συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρχει σύστημα ε, API, interface δηλαδή τυποποιημένο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε ούτε ε, πολλαπλά interface να υπάρχουν για κάθε χώρα και για κάθε τράπεζα, ούτε να είναι ε, επιλογή του καταναλωτή αυτό. Έτσι λοιπόν, εάν έχουμε ένα ανοιχτό τραπεζικό σύστημα με ε, ομαλές και τυποποιημένες κατά κάποιο τρόπο οργανωμένες συναλλαγές, μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Μέχρι στιγμής το πώς δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα. Κάποια στοιχεία κοινά στο σχέδιο της ε, ΕΤΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Interface είναι τα εξή. Εξ αρχής με την ε, ΕΤΑ έχει συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ειδικό Interface θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τον, παρόχο, για τον τρίτο πάροχο υπηρεσίας. Και οι οργανώσεις των καταναλωτών ήταν πολύ, ενδιαφε... Ε, ήταν πολύ ενθουσιώδεις. Fintech θεώρησε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο ή και αδύνατον να εξασφαλίσει καλό σύστημα πληρωμών και απαιτούσε πιο συγκεκριμένες διασφαλίσεις στις οποίες και εμείς εργαστήκαμε. Εργοδός η ΕΤΑ έκανε από πλευρά της τη δουλειά της. Η Επιτροπή είχε αμφιβολίες ως προς το αν θα μπορούσε ένα ειδικό interface να αντιμετωπίζει όλες τις πιθανές δυσκολίες και έτσι είπαμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε διαδικασίες και κίνητρα ε, για να περάσουμε στο interface το διατραπεζικό αλλά με πολύ συγκεκριμένους όρους μέσω των οποίων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτή η εναλλακτική. Βέβαια δεν υπάρχει αντιστοιχία όπως θα ήθελε η Fintech και οι τράπεζες ε, είπαν ότι θα είχαν ένα μηχανισμό που ε, θα τους επέτρεπε να καταλήξουν στο interface εάν έπρεπε να προσαρμόσουν ωστόσο το interface τους ούτως ή άλλως όπως το προτείνει η Fintex. Και προτείνουμε μία εξαίρεση για τις τράπεζες που έχουν το δικό τους interface και δεν είναι υποχρεωμένες να δώσουν τον εναλλακτικό μηχανισμό πέραν του ειδικού interface που διαθέτουν με σαφές κίνητρο προφανώς για τις τράπεζες να προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό σε καλό ειδικό interface και αν μέχρι εάν τρεις μήνες πριν από την θέση σε εφαρμογή του συστήματος έχουν αυτό καλό σύστημα, τότε οι εθνικές αρμόδες αρχές εξαιρούν τις τράπεζες αυτές υποχρεωτικά και έτσι αυτές οι τράπεζες δεν χρειάζεται να έχουν αναλλακτικό μηχανισμό. Και αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι τράπεζες δίνουν κάθε δυνατή έμφαση και προσπάθεια σε ένα καλό interface, ειδικό interface που να καλύπτει τις ανάγκες και των τραπεζών και της fintechs. Χιλιάδες τράπεζες λοιπόν που θα πρέπει να έχουν κοινέ προδιαγραφές για το interface αυτό, αντί κάθε μία να κάνει τις δικές επιλογές. Από τις ε, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα βλέπουμε ότι υπάρχει βούληση για μια καλή προσπάθεια και η Επιτροπή θα τις συνοδεύσει αυτές τις προσπάθειες για τις προδιαγραφές και βέβαια για την προστασία δεδομένων που απαιτείται. Επομένως, τεχνικές προδιαγραφές δεν θα έχουν πολύ λεπτομερή κατάλογο προϋποθέσεων για το interface, αλλά βασικούς κανόνες που θα επιτρέψει όλες τις δυνάμεις αγοράς να, ενώσουν, να ενωθούν για να, κάνουν, να ετοιμάσουν ένα καλό σύστημα προς όφελος του καταναλωτή αλλά και των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Um, Σας ευχαριστούμε. Φυσικά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Πάντως από τη δική μου σκοπιά έχουμε σημαντική πρόοδο. Γιατί δίνει τα κίνητρα στην ειδική διασύνδεση, ενώ προηγουμένως ήταν προσανατολισμένη στις ανεπιθύμητες συνέπειες. Δεν έχουμε ακόμη το κείμενο βέβαια. Θα ακούσουμε τον εισηγητή μας τώρα, τον Μάρκους Φέρμπερ. Ευχαριστώ πολύ. Και χαίρομαι που έχουμε πάλι τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε το, δεύτερη εκδοχή του Ισοδικίας για τις, ε, για τις υπηρεσίες πληρωμών, διότι τις τελευταίες εβδομάδες διαβάζουμε και στις γερμανικές εφημερίδες κάποια παράξενα για υπηρεσίες πληρωμών, υπηρεσίες πληροφοριών, λογαριασμού και ούτω καθεξής. Στις διαπραγματεύσεις ε, για το σύστημα πληρωμών για την PSD2, υπενθυμίζω το Κοινοβούλιο, ήθελε να έχει ένα σύστημα που να ισχύει στην Ευρωζώνη, που να επιτρέπει μια καλή ε, προστασία των ε, δικαιωμάτων του καταναλωτή και της, ε, και της ανάγκης βέβαια προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και βλέπουμε ότι η Google, το Facebook διαδίδουν ένα σενάριο τρόμου ότι θα πάρουν στα χέρια τους κάποιοι τα δεδομένα των τραπεζικών μας λογαριασμών. Λοιπόν, σπέβδω να πω ότι αυτό δεν ισχύει. Ωστόσο, προξένησε το, η διάδοση αυτού του σενάριου την ανάγκη για συζήτηση. Και η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών ε, προβληματίστηκε για το αν το PSD2 είναι σύμφωνο με, την, ε, με τον κανονισμό για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών. Φαντάζομαι ότι ισχύει αυτό, γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι παράνομο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα ήταν σκόπιμο και σε αυτό το χώρο συζητήσεων που βρισκόμαστε να πάρουμε επισήμως απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, και για να δούμε και τα μέληματα τα σχετικά με την προστασία του καταναλωτή, δεν αποφασίζει η τράπεζα εάν ε, είναι ικανοποιητικό ένα σύστημα πληρωμών, αλλά εγώ ως καταναλωτής, αν θέλω ε, να επιλέξω έναν αλλακτικό τρόπο πληρωμής, τότε θα πρέπει να μπορώ να το πράξω αυτό, χωρίς καθυστέρηση. Και έτσι θα ήθελα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, θα ήθελα να επισημανώ ότι είμαι ευγνώμων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το έθιξε, γιατί είναι κάτι που μας είχε απασχολήσει. Ωστόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ρωτήσω κάτι ακόμη να μας απαντήσει. Είναι τελικά οι εθνικές αρχές στο τέλος αυτής της διαδικασίας αρμόδιες για να δώσουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι και στα 28 κράτη-μέλη θα προβλέπεται αυτή η ποιότητα και ότι δεν θα βρεθούν στα μικρότερα ενδεχομένω ε, ή εκείνα τα οποία μπορεί να έχουν ένα πιο ανοιχτό σύστημα. Εν χωρίς να θέλω να καταδείξω κανέναν ένα σύστημα στο οποίο θα είναι πιο εύκολο να μην ε, προσφερθεί αυτή η δυνατότητα. Θα είναι για όλους ε, υπαρκτή η δυνατότητα οι αρχές οι εθνικές να επαληθεύουν ότι προσφέρονται οι δυνατότητες των πληρωμών για τον καταναλωτή. Και επίσης για τους μεγάλους πελάτες θα υπάρχει εξαίρεση σε σχέση με την με τα στοιχεία ταυτοποίησης του πελάτη. Το αγαπημένο παράδειγμα το ξέρετε, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν ε, οργανώνει ε, ταξίδια των υπαλλήλων της, δεν έχει τα προσωπικά δεδομένα του κάθε υπαλλήλου και τα στοιχεία του σε κάθε κράτηση και κάθε πληρωμή, ε, αλλά γίνονται αυτά στο όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα συνεχίσει αυτό ή θα πρέπει κάθε υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από εδώ και μπρος να ε, κάνει μόνο του την κράτησή του, γιατί διαφορετικά δεν θα του το επιτρέπει το σύστημα ταυτοποίησης μεγάλων πελετών. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα. Με την ε, με το Champions League, επί παραδείγματι. Τόσε ομάδες ταξιδεύουν κάθε τόσο. Η Bayern Μονάχου είναι σήμερα εδώ για να παίξει με το Anderlecht και προφανώς δεν ε, κλείνει εισιτήριο κάθε ποδοσφαιριστής για λογαριασμό του, αλλά η ομάδα για όλου. Ε, ταυτόχρονα όμως είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι αρχές του ε, συστήματο ταυτοποίηση του ισχυρού ή του μεγάλου πελάτη. Θα υπάρχει αυτό, θα δώσουμε μια περιοτεραιότητα μάλλον στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα γίνεται μια θα, θα, θα είναι δυνατό να συνεχιστεί μια σχετικά ομαλή δραστηριότητα οικονομική σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Σε αυτό θα ήθελα απαντήσεις. Thank you. Σας ευχαριστώ. Θα ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα έχουμε πρώτα ένα γύρω ερωτήσεων από την Ομιγύρη και μετά θα δώσω το λόγο στους προσώπους της ΕΚΤ και της ΕΑΤ. Ο κύριος Λούντβικσον από τους συναδέλφους. Πρώτα Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος. Θα ήθελα να ρωτήσω για την ε, παροχή υπηρεσιών από 33 τρίτον. 33-32-93 υπηρεσία των υπηρεσιών και οι προδιαγραφές που προβλέπει περιγράφουν τις υπηρεσίες, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ε, υπηρεσιών που είναι υποχρεωτικό να είναι ουδέτερες. Έτσι ώστε να εξασφαλίζεται και επίπεδο ισότιμο ανταγωνισμό στην αγορά των πληρωμών. Και πρέπει ταυτόχρονα να αρχίσουμε σιγά σιγά να βγαίνουμε από το σύστημα το οποίο χρησιμοποιούνταν τα τελευταία 15 χρόνια. Θα υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα για μία τράπεζα να εισάγει εξαιρέσεις θα είναι εγγυημένη η αρχή της πρόσβασης στην τράπεζα για τον πελάτη ή θα υπάρχει δυνατότητα να αποκλειστούν κάποιοι πελάτες fintech από τις μεγάλες τράπεζες. Θα δώσουμε έμφαση δηλαδή στον ε, θεμητό ανταγωνισμό, στις ισότιμες ε, συνθήκες ανταγωνισμού. Ελπίζω να μπορέσει να απαντήσει η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Uh, Πρώτα να δούμε ε, ποιοι συντονιστέ είναι στην αίθουσα και μετά θα περάσουμε στο Catch the Eye. Catch the Eye και εγώ και ο κύριος Χέις, η κυρία Μπέρες, ο κύριος Χέις. Ευχαριστώ. Και εκτιμώ τα σχόλια των συναδέλφων για το θέμα αυτό. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε τελικό στάδιο της διεκπαιρέωσης αυτού του ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου. Έχουμε εκδηλώσει εδώ και πολύ καιρό ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η ειδική διασύνδεση, το Dedicated Interface, είναι καλύτερος τρόπος για να εμπλέξουμε τις τράπεζες στην ανάπτυξη των APIs και φυσικά με πανευρωπαϊκές προδιαγραφές. Βέβαια, αν τελικά έχουμε και μια εναλλακτική λύση για το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο, ε, υπάρχει κίνδυνος ε, σοβαρού κατακαιρματισμού της αγοράς που απευχόμαστε φυσικά και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό το κίνδυνο, το να απαιτήσουμε από τις τράπεζες ταυτόχρονα να εφαρμόσουν μια τέτοια ε, δεύτερη λύση εναλλακτική όταν ήδη προσπαθούν να θεσπίσουν μια ειδική διασύνδεση, ένα dedicated interface, σε αποτρεπτικά όταν προσπαθούν να καταλήξουν σε μια κοινή προδιαγραφή για το dedicated interface. Βέβαια έχουμε την Τραπεζική Ένωση, θα μου πείτε, και θα ίσως θέλουμε ενιαίες προδιαγραφές για τις τραπεζικές ε, δραστηριότητες, στο μέτρο του δυνατού. Μια, ένα εύρυθμο, μια εύρυθμη ειδική διασύνδεση, ένα εύρυθμο dedicated interface θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε ασφάλεια των δεδομένων. Και ε, η άλλη μέθοδος δεν εξασφαλίζει στους καταναλωτές το ίδιο επίπεδο ασφάλειας, γιατί ε, Τη παροχή θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για την υπηρεσία που παρέχουν. Αν λοιπόν αναπτύξουμε ένα dedicated interface, μια ειδική διασύνδεση που θα εφαρμόζεται ad hoc και για τέτοια fallback μέτρα, ε, νομίζω ότι δεν θα υλοποιήσουμε τον ε, επιδιωκόμενο μας στόχο. Θα πρέπει ε, να λάβουμε σοβαρά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο, το RTS. Και αν ε, επιβάλλουμε ένα τέτοιο, μια τέτοια απέτηση ε, σε σχέση με, τη, με το API, στη δεύτερη, στο άρθρο 97 της ε, δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών, ίσως έχουμε αντίθετο αποτέλεσμα. Περιμένω την, το σχολιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Υπερβάσου Μπερές. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε και για τη δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών αυτή τη συζήτηση ελέγχου, γιατί εδώ και καιρό ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και θα πρέπει να κάνουμε πιο νυφάλια συζήτηση, προκειμένου να βρούμε μία απτή λύση για να επιτρέψουμε και τον, τη συνύπαρξη του ανταγωνισμού με την ασφάλεια η ύπαρξη τεχνολογιών API είναι η κατάλληλη λύση, γιατί συνδυάζει τη, τη σύγχρονη εποχή με την ασφάλεια. Τώρα το fallback option. Αν δεν γίνει σωστή πλαισίωση αυτής της πιθανότητας της ε, μετάπτωσης λειτουργίας, ίσως ε, διονυστεί η σημερινή κατάσταση και δεν είναι η επιθυμητή λύση, δεν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα το fallback σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες των ε, fintech. Αντιλαμβανόμαστε τις ανησυχίες τους και την μεριμνά τους υπέρ της ανάπτυξης και ανατομίας, αλλά θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους μας να ε, νομοθετούμε χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο, χωρίς να το έχουμε θωρακίσει. Και από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή αυτό το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο, θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να μπορούν να εξακριβώνουν τη σωστή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, γιατί εδράζεται σε μια συμφωνία εμπιστοσύνης, είτε εκ μέρους των τραπεζών, είτε των FinTech. Για αυτή την ερώτηση θα πρέπει να θέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέραν του ρυθμιστικού τεχνικού προτύπου του RTS, πώς θα εξασφαλιστεί ο έλεγχος και η εποπτεία της, θέσης, της ουσιαστικής θέσης εφαρμογής αυτής της λεπτής ισορροπίας που προτείνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Έχω και εγώ κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις και φυσικά μας ενδιαφέρουν και οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Α, από ό,τι κατάλαβα, το κρίσιμο θέμα για αξιολόγηση είναι αυτό το θέμα της εξαίρεσης, γιατί ε, ο μηχανισμός ειδική διασύνδεσης ε, θα πρέπει να διευκρινιστεί. Πώς ε, θα τηρηθεί αυτή η υποχρέωση ακριβώς ταυτότητας 66 Δέλτα και 67 που αναφέρονται στη δεύτερη οδηγία και την πρόβλεψη το τρίτο μέρος να έχει πρόσβαση μόνο στις ε, πληροφορίες που χρειάζεται για να παράσχει την απαιτούμενη υπηρεσία. Φαντάζομαι εσείς θα μας τα εξηγήσετε καλύτερα σε οποιαδήποτε επιλογή, γιατί υπάρχει δυνατότητα μετά το λειτουργίας του fallback. Οπότε πώς θα αποφευθεί αυτός ο κίνδυνος να παραβιαστεί η απέτηση η νομοθετική. Και το θέμα είναι οι εξαιρέσεις. Πώς εξαιρέσεις από το fallback θα εφαρμοστούν. Ε, από ό,τι κατάλαβα, η αρμόδια αρχή θα χορηγεί την εξαίρεση υπό την προϋπόθεση της στήρησης των όρων. Καταρχήν, είναι επαρκής οι προϋποθέσεις ώστε να έχουμε μια υψηλών προδιαγραφών ειδική διασύνδεση, dedicated interface, και να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτό το dedicated interface οι τράπεζες και να έχουν τον απαραίτητο χρόνο ώστε να μην μπουν στον πειρασμό να πέσουν στο fallback που ίσως φέρει ανεπιθύμητες συνέπειες. Ε, τι γίνεται με την απόσυρση της εξαίρεσης. Είναι εξάντε ο μηχανισμός εκ των προτέρων ή θα ουσιαστικά έχουμε de facto υποχρέωση εφαρμογής του fallback. Έχουμε δηλαδή επαρκείς διασφαλίσεις και μηχανισμούς ώστε να δημιουργήσουμε κίνητρα και να καταλήξουμε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ώστε να έχουμε φαινός άνοιγμα, ανταγωνισμό, αλλά ταυτόχρονα και ασφάλεια με ένα τέτοιο dedicated interface μεταξύ των τραπεζών, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, αυτή η ειδική διασύνδεση. Ο μηχανισμός είναι σχεδιασμένος ε, με τέτοιο τρόπο ώστε να μας επιτρέψει την υλοποίηση του στόχου και να λειτουργήσει πραγματικά. Μας ενδιαφέρει λοιπόν και η άποψη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που φαντάζομαι θα μα πει ότι ναι, λειτουργεί το σύστημα, αλλά μα ενδιαφέρουν και οι απόψει τη ΕΚΤ και τη Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Ευχαριστώ για αυτά τα σχόλια. Να ξεκινήσω με το θέμα του ε, μηχανισμού δεύτερης λύσης, fallback mechanism, σε περιπτώσει πολλοί θεωρούν ότι θα είναι μια εύκολη επιλογή. Να περάσει κάποιος δηλαδή σε αυτήν την δεύτερη επιλογή όταν υπάρχει. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Εμείς δεχτήκαμε απολύτως την πρόταση της EBA να είναι υποχρεωτικό να περάσει κανείς από το dedicated interface όταν υπάρχει. Βεβαίως θα πρέπει να είναι αρκετά καλό αυτό το interface. Ελπίζουμε να είναι τόσο καλό και δοκιμασμένο που η απέτηση να υπάρχει ένας μηχανισμός ε, ε δεύτερης επιλογής ε, κάποια στιγμή να αρθεί. Αυτό θα προτιμούσαμε όλοι. Θέλουμε όλοι να περνάμε από το NPI ως μηχανισμό πρόσβασης. Δεν, αποφασίσαμε πάντως να απαγορεύσουμε αυτή, αυτή την πρακτική. Αν μια τράπεζα επιλέξει αυτή την οδό μπορούμε, μπορούμε να το δεχτούμε. Δηλαδή προβλέπεται από την νομοθεσία. Εμείς απλώς είπαμε ότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν στην fintech μια, ένα συγκεκριμένο interface. Διότι όταν υπάρχει αυτό το ε, interface είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή πιέσαμε κάπως το PST2 στα όρια του για να μπορέσουμε να επιταχύνουμε μέσω της διαδικασίας αυτής τη μετάβαση προς ε, ε, τυποποιημένη πανευρωπαϊκή πανευρωπαϊκό τυποποιημένο interface, dedicated interface. Τώρα πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια συνεπή εφαρμογή δηλαδή ε, αυτής της εξαίρεσης. Εμείς προβλέπουμε πριν χορηγηθεί η εξαίρεση από μια εθνική αρμόδια αρχή να πρέπει να έχετε σε επαφή με την EBA έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια συνέπεια Υπάρχει και έλεγχος από τις ίδιες κεφαλαίες αγορές, εφόσον αυτό το dedicated interface έχει οδηγήσει σε μία εξαίρεση, αλλά δεν λειτουργεί για τους ε, παρόχους ε, τρίτων. Ε, και αυτοί μπορούν βεβαίως, τους τρίτους παρόχους, αυτοί μπορούν να ε, διαμαρτυρηθούν στην περίπτωση αυτή και πρέπει οι εθνικές αμμόδιες αρχές να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις προβλέπονται στο PSD2, αυτό θα το εξασφαλίζει η Κομισιόν, αλλά και ε, τα τεχνικά πρότυπα η εξαίρεση δηλαδή μπορεί να χορηγηθεί μόνο εφόσον είναι, είναι ικανοποιημένη η κεφαλαία αγορά. Αυτό που θέλουμε είναι οι κεφαλαία αγορές να συνεργαστούν για τα πρότυπα API, ε, για πρότυπα API που θα λειτουργούν και για τις δύο πλευρές. Το θέμα της προστασίας των δεδομένων τώρα. Ε, βεβαίως ε, είναι αντικείμενο αντιπαράθεσης, έχουμε εργαστεί σκληρά επ' αυτού έγινε και ένα εργαστήρι για την εφαρμογή με τα κράτη-μέλη όπου εξετάσαμε και οι επιπτώσεις του GDPR ε, για τις διαδικασίες που θα πρέπει να θεσπιστούν έτσι ώστε να λειτουργήσει το PST2. Υπάρχουν λύσεις πάντως. Ε, το εξετάσαμε αυτό και με την νομική υπηρεσία. Υπάρχουν, ε, υπάρχει μια φάση που να επιτρέπει τη διαβάση δεδομένων μεταξύ τραπεζών και, παρόχων, και τρίτων παρόχων. Αυτό θα πρέπει να γίνει βεβαίως με την πλήρη ε, συνένεση και σε πλήρη διαφάνεια, πλήρη συνένεση των χρηστών. Όποιος δεν θέλει να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια υπηρεσία ε, δεν πρόκειται να δευαστούν τα δεδομένα του. Ε, υπάρχει πολύ μεγάλη πρόοδο δηλαδή σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση, γιατί αυτή τη στιγμή με το GDPR προβλέπονται πρόστιμα. δηλαδή κινδυνεύει να χάσει την άδειά του ε, ο φορέας εάν δεν ε, σεβαστεί τις διατάξεις, τις απαιτήσεις του PST2. Δεν μπορούν να αντιδρύσουν τα δεδομένα αυτά για πάντα και να τα διαβάζουν όπως θέλουν. Το τελευταίο που ήθελα να πω έχει να κάνει με τις πληρωμές ε, των επιχειρήσεων corporate payments. Είχαμε συζητήσει μια πρόταση για μια παρέκκληση σε ό,τι αφορά τα corporate payments. Το θέμα λοιπόν που έθεσε ο κ. Φάβα έχει λυθεί. Ξέχασα όμως κάτι ακόμα. Το Η ελεγχόμενη πρόσβαση σε πληροφορίες ταυτοποίησης των TPPs. Αυτό θα προτελέσει αντικείμενο περαιτέρω εργασιών σε άλλη νομοθεσία επίπεδου 2, δηλαδή level 2. Ίσως ο συνάδελφος του EBA μπορεί να πει κάτι από αυτού. Ναι, και η απέτηση ταυτοποίησης καλύπτεται και αυτή από το IPS. Ναι, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ που μου δώσατε ε, χρόνο ε, να παρέμβω εδώ. Χαίρομαι ε, που βρίσκομαι εδώ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η BA αυτή που ελέγχει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι ευχάριστο για μας. Είναι καλύτερο να σχολιάζει κανείς από το να κατηγορείται. Εμείς εδώ και δύο χρόνια ερχόμαστε από αυτού του συστήματος. Φαντάζομαι ότι όλοι εδώ ενδιαφέρεστε έτσι ώστε να υπάρξει επιτυχία με αυτό το RDS. Είμαστε μόλις 6 μήνες από την εφαρμογή του PST2. Έτσι λοιπόν σε επίπεδο μελών ε, υπάρχει ετοιμότητα, ε, λαμβάνει η χώρα, λαμβάνει χώρα ήδη επεξεργασία ε, αιτήσεων για να μπορέσουν να αρχίσουν να παρέχουν παράγοντες υπηρεσίε από την Ιανουάριο και μετά. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα ακόμα βήμα. Δεν έχουμε δει ακόμα βέβαια το κείμενο, οπότε είναι δύσκολο να αξιολογήσουμε τις τροποποιήσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι ο διάβολος κρύβει τις λεπτομέρειες ως γνωστόν, να αναφερθώ σε δύο-τρία σημεία όμως που ανέφερε μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εισαγωγή αλλά και πριν από λίγο. Αν καταλάβαμε καλά, θα υπάρξει μια εξαίρεση σε ό,τι αφορά αυτή την δεύτερη επιλογή, το fallback option. Αυτό πάει προς σωστή κατεύθυνση, διότι όπως ξέρετε η EBA είχε πολύ σημαντικές επιφυλάξεις απέναντι σε αυτήν την ιδέα της δεύτερης επιλογής. Θεωρούμε ότι αυτό δίνει αντικίνητρα ε, και μπορεί να υπονομεύσει την δημιουργία APIs ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξαίρεση αυτή λοιπόν πάει προς σωστή κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει να δούμε το ακριβές κείμενο, διότι αν καταλάβαμε καλά οι εθνικές αρχές είναι αυτές που θα πρέπει να αποφασίσουν κατά πόσο αυτή η εξαίρεση θα χορηγηθεί ή όχι. Και αυτό δημιουργεί δύο ζητήματα. Πρώτον, το βάρος της συμμόρφωσης περνάει από το από την, ε, τον φορέα τον οικονομικό προς την ε, Εθνική Αρχή. Ε, και δεν είναι αυτό αυτός τρόπος λειτουργίας για τον, για τον, για τον κανονισμό μας, γιατί ο βάρος τελικά τον αναλαμβάνει η Εθνική Αρχή για την χορήγηση αυτής της εξαίρεσης με τον σωστό τρόπο και με τρόπο που να επιτρέπει στην αγορά να λειτουργήσει. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε λεπτομερώς πώς θα λειτουργήσει αυτό. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο είναι ο ρόλος της EBA στη διαδικασία αυτή. Αν κατάλαβα καλά, ε, η Εθνική Αρχή θα πρέπει να συμβουλευτεί την EBA για τη χορήγηση της εξαίρεσης. Ε, εμείς συμφωνούμε βεβαίως ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια σε επίπεδο Ένωσης για το πώς θα χορηγούνται αυτές οι εξαιρέσεις. Ο ρόλος της EBA λοιπόν ε, εκ πρώτης εδώ λογικός μας φαίνεται αλλά τι σημαίνει consult with EBA, e να, συμβουλ, να διαβουλευτεί, να συμβουλευτεί την EBA. Έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε κάτι εμείς, να επιβάλλουμε κάτι, αν δεν κάνει κάποια πράγματα η Εθνική Αρχή όπως ε, ε, πρέπει, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Επίσης, η εξαίρεση της αξιολόγησης, ε, του κατά πόσο να χορηγηθεί μια εξαίρεση ή όχι, θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Πρέπει να προσέξουμε τι, τι εξετάζεται το, το στοιχείο, το, το, η πτυχή της ασφάλειας ε, του RDS. Αυτό όντω πάνω το κάνει η Εθνική Αρχή και η EBA, αν και είναι σημαντικό το διοικητικό αυτό. Πρέπει να δούμε αν οι εθνικές αρχές έχουν επαρκεί πόρου, ε, σε προσωπικό δηλαδή εννοώ, σε ανθρώπινου πόρου, ε, διότι μπορεί να έχουμε ένα σημαντικό αριθμό APIs προς αξιολόγηση. Αυτό που είναι κρίσιμο όμως είναι τι ακριβώς θα αξιολογηθεί. Μόνο το, η πτυχή που αφορά την ασφάλεια ή οι ανησυχίε του TPP, διότι το TPP δεν έχει πρόβλημα με την ασφάλεια, είναι ότι μπορεί να μην είναι το interface αξιόπιστο ή μπορεί να, είναι, να μην είναι διαθέσιμο σύν χρόνο. Ε, τι θα μπορεί να αξιολογήσει η Εθνική Αρχή, την, ε, θα μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσο θα υπάρχει διαθεσιμότητα σε τεχνικό επίπεδο θα υπάρχει πραγματογνωμοσύνη απαραίτητη όμως από το προσωπικό για να γίνει η, θα υπάρχουν δεξιότητες στα προσόντα ε, για να αξιολογηθεί τεχνικά αυτό το interface. Η EPA πάντως δεσμεύεται να είναι στη διάθεσή σας το ερχόμενο έτος και προς τα TPPs και προς τις τράπεζες για να δημιουργηθούν αυτά τα APIs και αναμένουμε να δούμε ε, Γραπτό, βεβαίω και τι ιδέε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ρόλο του CBA στη διαδικασία αυτή και θα δούμε. Καλό θα ήταν πάντως να υπάρξει μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί τον Μάιο-Ιούνιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι καλό ότι θα ζητηθεί άποψη τη EBA διότι η αξιολόγηση αυτή ε, της, ε, των εξαιρέσεων, η ε, η αντιστροφή του βάρους ε, της ε, συμμόρφωσης είναι μια σημαντική υπόθεση. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέσσερα στο σχόλια. Πρώτον, ότι σεβόμαστε την νομοθετική διαδικασία και πρέπει να δούμε τι θα προκύψει από αυτήν. Δεύτερον, ευπρόσδεκτη η τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί το στόχο της ανανέωσης ε, της καινοτομίας και του ανταγωνισμού. Τρίτον, ευπρόσδεκτη η τροποποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γιατί θεωρούμε ότι συνιστά κίνητρο ώστε οι τράπεζες, οι και γενικά οι παράγοντες στην αγορά να αναζητήσουν συνένεση στην πράξη για τους πρακτικούς όρους τους απαραίτητους που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ενοποιημένης αγοράς για να το πω διαφορετικά για να διευκρινιστούν οι πρακτικές συνθήκες υπό τις οποίες η API θα είναι καλή και πρέπει να δούμε βεβαίως σε ποιο βαθμό μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσει με τη συμφωνία αυτή η αγορά σε τυποποιημένα interface. Αυτό μένει να το δούμε. Είναι απαραίτητο τεχνικά το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά τα πάντα θα κρυθούν από το πόσο διατεθειμένη είναι η αγορά και οι παράγοντες, οι συντελεστές, ώστε να συμφωνήσουν σε συγκεκριμένους όρους για ένα καλό API. σε σχέση με τη δική μας την αρχή και το σώμα πληρωμών λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο προσδορίζει καλές προϋποθέσεις, έχει σημειώσει καλή πρόοδο. Δεν έχουμε φτάσει στο πέρας. Και βεβαίως ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει το έργο των συντελεστών της αγοράς για την επίτευξη καλών όρων. Ο κύριος Φόξ δεν είναι εδώ για την επόμενη ερώτηση, αλλά κατά εξαίρεση θα σας διαβάσω το σχόλιο. Ίσως και ο Μάρκος θα θελήσει να επανέλθει, ίσως και η Επιτροπή. Πρώτα όμως ας προβώ στην ανάγνωση. Ο κύριος Φόξ θα προτιμούσε να έχει ένα αντίγραφο του ελληνικού κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως άλλωστε και εμείς. Τρεις ερωτήσεις ακολουθούν, γιατί η Επιτροπή προχωρεί στην επιλογή fallback option plus, ε, δηλαδή της εναλλακτική λύσης. Δεν φαίνεται αυτό να ενισχύει το σύστημα. Τυποποιημένο MPI θα ήταν πιο αποτελεσματικό μέτρο για την ε, προαγωγή των σχέσεων μεταξύ των τραπεζών και των πελατών, γιατί πρέπει να υπάρχουν 150 ευρώ και 5 συναλλαγές σωρευτικά πριν πριν είναι υποχρεωτική μετάβαση στο σύστημα. standards required not, to not have in place a fallback. Please can they explain how they will ensure that banks continue to meet these requirements? So these were requests from Mr. Fox and Marcus, please. Ο κύριος Γουαλτιέρο ολοκλήρωσε την ανάγνωση του κειμένου και δίνει το λόγο στον κύριο Φέρμπερ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις ε, απαντήσεις που δώσατε στις δικές μου ερωτήσεις. Δεν το είχατε πράξει την προηγούμενη φορά. Σημαντική βελτίωση. EBA, ACT, Επιτροπή. Φαίνεται ότι δεν είχαν σωνηθεί πιο πριν. Βλέπουμε μεγάλες αντιφάσεις ε, που και εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε πριν δούμε το κείμενο στις λεπτομέρειές του. Ίσως μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για το χρονοδιάγραμμα. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά, αλλά αν δεν είναι ικανοποιημένη η ΕΤΑ για το χρονοδιάγραμμα ή δεν γνωρίζει η αγορά. Και πρέπει να πούμε ότι όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται για το green scraping και τα λοιπά ε, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει δυνατότητα όσο δεν έχει μπει σε λειτουργία το ΕΡΤΕΣ Είναι πολύ έσπιστος δυνατότητες από ότι μετά τη θέση εφαρμογή. Γι' αυτό λοιπόν ε, να ξέρουν αυτοί οι οποίοι καθυστερούν ότι θα έχουμε περιορισ... πιο περιορισμένη προστασία προσωπικών δεδομένων και καταναλωτών όσο δεν έχει προχωρήσει η δεύτερη οδηγία, το PSD2 δηλαδή, για να κλείσουν τα, τα κενά και τα παραθυράκια. Και επίσης η Επιτροπή, η ΕΚΤ, κάποιος τους παντοχτές, έκανε μια ανακοίνωση ότι άρχισαν οι instant payments, στιγμιές πληρωμές, δηλαδή εμβάσματα ε, που διαρκούν ένα δευτερόλεπτο και όχι μία μέρα. Διερωτώ με, μήπως έχουμε εμπλακεί σε μια συζήτηση που ανοίξει στο παρελθόν, όταν πια έχουν ε, ήδη εγκαθιδρυθεί άλλες μέθοδοι πληρωμών στους οποίες δεν χρειάζομαι κανέναν διαμεσολαβητή εγώ ως κάτοχος ενός λογαριασμού δηλαδή μπορώ και χωρίς ανάγκη από τράπεζα, από επιστοτική κάρτα, από έντυπο εμβάσματος να στείλω λεφτά κάπου. Μήπως λοιπόν μιλούμε για άσχετα θέματα πλέον. Έπρεπε να το πω και αυτό γιατί είναι τέτοιες οι δυνατότητες ε, που μας, ε, με τις οποίες μας πλημμυρίζει ο ψηφιοποιημένος κόσμος, που στις τεχνικές προδιαγραφές μας είναι πολύ πίσω. Ε, οι τελικές παρατηρήσεις επιτροπής τώρα δεν έχει απαντηθεί εκτενώς η ερώτησή μου για το πώς η εξαίρεση του fallback εφαρμόζεται πρακτικά ως ε, η κύρια επιλογή και ποιες είναι ε, οι προϋποθέσεις για την ε, άρση των κυρώσεων και πώς θα αποφύγουμε τον, την αντιπαλότητα μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά δυσκολεύοντας ιδιαίτερα την εφαρμογή αυτής της εναλλακτικής λύσης και αυτό που είπε φυσικά ο συγκητής είναι πολύ σημαντικό το θέμα, το χρονικό δηλαδή. Να ξεκινήσουμε από το χρονικό ζήτημα. Στις 27 Νοεμβρίου περιμένουμε την ε, υιοθέτηση της πρότασης. Θα δημοσιευθεί τότε το έγγραφο σε όλες τις μεταφράσεις. Οπότε μπορείτε αμέσως κι εσείς ε, να ξεκινήσετε την επεξεργασία δικαιούστε ένα τρίμηνο, αν δεν το εξαντλήσετε, ακόμη καλύτερο. Πάντω αντιλαμβανόμαστε ότι θέλετε να το εξετάσετε ενδελεχώ. Ό,τι αφορά τι εξαιρέσει από τι απαιτήσει ε, για την εναλλακτική λύση, το fallback, ε, εμεί πιστεύουμε ότι αν οι τρίτοι πάροχοι, οι TPPs, μπορούν ε, μέσω του online interface των τραπεζών να το κάνουν και μέσω του, της ειδικής Είναι υποκατάστατο αν οι τράπεζες προβλέπουν διασυνδέσεις που επιτρέπουν στους τρίτους παρόχους να εργάζονται, να δουλεύουν μέσω του, της ειδική διασύνδεσης, δεν χρειάζεται να περνάνε στο, το online ε, interface. Αν όμως η κατάσταση επιδεινωθεί και αν ε, καταστεί αδύνατο κάτι τέτοιο, όπως συνέβη στο παρελθόν, τότε οι εθνικές ε, αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αποσύρουν την ε, εξαίρεση, να την ανακαλέσουν και μέσα σε δύο εβδομάδες, ε, έχουν δύο εβδομάδες για να ανακαλέσουν την εξαίρεση και τότε οι τράπεζες θα πρέπει να επαναφέρουν ένα εύρυθμο API, μια εύρυθμη διασύνδεση προγράμματος εφαρμογών ή να ε, ενσωματώσουν τον εναλλακτικό μηχανισμό, το μηχανισμό fallback. Τώρα, γιατί προτείναμε το Fallback Plus, τον ενισχυμένο αναλλακτικό μηχανισμό, ρώτησε ο κύριος Φόξ. Η ιδέα μας ήταν ότι αν ο, δεν υπήρχε ο μηχανισμός ο εναλλακτικός, γιατί μια τράπεζα έχει τυχή εξαίρεση και δεν σε αυτή η ειδική διασύνδεση, το Dedicated Interface, μέχρι όταν αποκατασταθεί κάποιο εύρυθμο interface θα πρέπει να έχουμε μια διάμεση λύση. Και με βάση το άρθρο 115.5 Τη δεύτερη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών ε, επιτρέπουμε στον τρίτο πάροχο, στον TPP, να χρησιμοποιήσει το online banking interface με ταυτοποίησή του και ενημέρωση των ρυθμιστικών αρχών και της ενδιαφερόμενης τράπεζας για την έκτακτη αυτή διαδικασία. Ε, εξακολουθεί να είναι έκτακτη αυτή η διαδικασία και να πόκεται στη διακριτική ευχαίρεια των τραπεζών πλήρως να αποτρέψουν τέτοια φαινόμενα. Δεν θέλουμε screen scrapping αλλά επαφιόμαστε στις τράπεζες, στη συνεργασία τους ό,τι αφορά την ενσωμάτωση τέτοιων interface και την αποτροπή τέτοιων φαινομένων. Μάλιστα. Έχουμε και 10 λεπτά ακόμη που πρέπει να αφιερώσουμε στο δεύτερο θέμα. Το ρύθμιση τεχνητού, τεχνη, τεχνητού προτύπου για τις ε, συναλλαγές στα πλαίσια του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, IFR. Έχουμε το κείμενο. Δεν ξέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει να κάνει κάποια σχόλια. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ λακωνική. Θα ήθελα απλώ να υπογραμμίσω ότι έγινε η πρώτη συνεδρίαση ελέγχου στις 22 Ιουνίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κείμενο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Οκτωβρίου, ένα κείμενο που ευθυγραμμίζεται πλήρως ε, με, με το αποτέλεσμα της συζήτησης. Θέλουμε ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που θα εφαρμόζουν τον, ε, την απέτηση του κανονισμού για ε, κάρτες πληρωμών και, και τους ε, παρόχους και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ανταγωνισμό και σε αυτό το σύστημα πληρωμής με κάρτες που μέχρι στιγμής ήταν ε, το πιο δαπανηρό στην πράξη. Στόχος λοιπόν είναι να αποφύγουμε ε, κατακόρυφα ε, ολοκληρωμένες ε, ε συστήματα πληρωμών και να ευνοεί τους δικούς τους παρόχους. Θέλουμε μια λειτουργική, ένα λειτουργικό διαχωρισμό των συστημάτων συναλλαγών με κάρτες και των οντοτήτων παροχών. Τώρα η οι ε, πελάτες μπορούν πολύ εύκολα να χρησιμοποιούν τις οντότητες για τις συναλλαγές με κάρτες. Ενώ στον κλάδο οι, ευρωπαϊκές, οι ευρωπαϊκοί φορείς ήδη έχουν εφαρμόσει κάποιο βαθμό διαχωρισμού. Και αυτό που θα κάνει και θα βοηθήσει το ρυθμιστικό τεχνικό πρότυπο είναι να εξασφαλίσει μια εναρμονισμένη προσέγγιση σε όλο τον κλάδο. Και επίσης προσθέτει και την εποπτεία από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην όλη διαδικασία. Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε απορίες και το συ... περιμένουμε τη συμφωνία από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να τεθεί σε εφαρμογή και εμπράκτος η νέα πρόταση από τον Ιανουάριο. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, θα είμαι στον πιο σύντομος θα κάνω μια συζήτηση για το θέμα βέβαια της πολιτικής ε, τάξης και της διάκρισης ε, στην οποία των, των διαχωρισμών που θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των πλευρών και για να αναφερθώ στη τελευταία παρατήρηση η πολύ αυστηρή ερμηνεία του δικαίου του ανταγωνισμού και έχουμε να κάνουμε την ε, Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στην τελευταία ανάλυση εδώ. τελικά οδηγεί στο να υπάρχουν ε, μόνο δύο συστήματα πιστοτικών καρτών που μπορούν να εξυπηρετηθούν, να εξυπηρετήσουν το σύστημα, δηλαδή οι δύο μεγαλύτερες και μήπως τελικά τα λοιπά συστήματα πέφτουν εκτός ε, του συστήματος. Αυτές ήταν οι προκατακτικές μου παρατηρήσεις και ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Άρλη, συνάδελφε. Παρακαλώ. Ναι, πρόεδρε. Συμφωνώ με την ε, πρόταση της Επιτροπής στο διαχωρισμό των συστημάτων ε, πληρωμών πιστοτικών κρατών και της ε, εξεργασίας των στοιχείων. Άλλωστε ορίζεται και στην νομοθεσία ότι θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη ε, τα συστήματα πληρωμής από την οργάνωση. Χαίρομαι λοιπόν που έχει καταθέσει την πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περισσότερο ανταγωνισμό, περισσότερη αγορά και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς. Λοιπόν, εφόσον δεν θέλει κάποιος άλλος το λόγο, ναι. που να θέλει το λόγο για το πράξη και εξοδότηση, Φαντάζομαι δεν έχει κάποιος κάποια αντίρρηση. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θέλει να πει κάτι. Ναι, επειδή τέθηκαν κάποια ερωτήματα. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε για να απαντήσω στον κύριο Φερ Βέρμπερ. Ε, είπε ότι με μια αυστηρή ε, ότι χρειάζεται μια αυστηρή ε, ερμηνεία των κανόνων ανταγωνισμού και τι συμβαίνει ε, με τα συστήματα αυτά, με τις κάρτες, πληρωμές με κάρτα. Ε, όταν έγινε η μελέτη αντικτύπου, εξετάσαμε ποια είναι η κατάσταση στην αγορά και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ήδη είχαν, κάνει, είχαν πάρει πρωτοβουλία αυτορύθμισης στο σύστημα πληρωμών ΣΕΠΑ ήδη, οπότε υπήρχε ήδη ένας διαχωρισμός αυτό που θα επηρεαστεί δηλαδή κυρίως είναι τα μεγάλα διεθνή ε, προγράμματα που δεν έχουν εφαρμόσει ε, σε αυτό το βαθμό αυτή την αρχή της ανεξαρτησίας και βεβαίως οι ε, ρυθμιστικές αρχές οι εθνικές είναι ήδη σε επαφή με αυτά τα προγράμματα, συστήματα καρτών και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. σίγουρα ε, δεν θα δυσκολεύσουν, τα πράγματα για τα ευρωπαϊκά συστήματα διότι εκεί ήδη έχει γίνει η προσαρμογή τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει μια κάποια, ένας κάποιος διαχωρισμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε ε, αυτό το κομμάτι της συνεδρίασης. Ε, θα διαβάσουμε προσεκτικά το κείμενο για το RDS που θα υποβληθεί ε, στο τέλη του 2017 στις 27 μάλλον του μήνα ε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά σίγουρα πάντως πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα διότι έρχεται να αντιμετωπίσει μια σειρά από ανησυχίες ε, απολύτως βάσιμες. Ε, ευχαριστούμε την ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την EBA, την Κομισιόν, την παρουσία τους εδώ. Κάναμε την αξιολόγηση και τώρα να περάσουμε στην ψηφοφορία. Χρειάζομαι βέβαια στον κατάλογο κατάλογο. Λοιπόν, μια στιγμή. Μια στιγμή. Και θα αρχίσουμε σε λίγο τη ψηφοφορία. Meanwhile, let's have a test. A test. Εν τω μεταξύ, κάνουμε μια δοκιμή. Δοκιμαστική ψηφοφορία. Okay. So we Ωραία. Ήφρεσε νέα. Επανέρχεται στην Επιτροπή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή για την ταχύτητα στην διεκπαιρέωση ονομαστικά και ψηφίζουμε. Vote is closed. Πέρας. 38 υπέρ 12 κατά, μία αποχή και εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Δεύτερη ψηφοφορία σε άλλο θέμα πάλι fast track. Ταχείας διαδικασίας. Η ιεράρχηση των μη εξασφαλισμένων πιστωτών σε περίπτωση πτώχευσης και πάλι συγχαρητήρια για την ταχύτατη διεκπαιρέωση των διαπραγματεύσεων και αρχής ψηφοφορία. Vote is closed. 44 8 κατά. Αποχές 0. Εγκρίνεται το κείμενο και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Σχέδιο εκθέσεως Χώνος Φερνάντες, ετήσια έκθεση ΕΚΤ 2016. Περβός. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Λυπούμε ιδιαίτερως εδώ που ομάδες που έλαβαν μέρος στην επεξεργασία των συμβαστικών προτάσεων μέχρι και τελευταία στιγμή εν τέλει ξαναζητούν χωριστή ψηφοφορία για πολλές τροπολογίες τους που στην πραγματικότητα όμως καλύπτονται από τις συμβαστικές γιατί υποτίθεται ότι συμβάλλουμε στις συμβαστικές και μετά επαναφέρουμε τις τροπολογίες μας. Η δική μας ομάδα θα απόσχει στις τροπολογίες αυτές για τις οποίες τελευταία στιγμή ζητήθηκε χωριστή ψηφοφορία κατά παράβαση του πνεύματος του συμβασμού και των συμβαστικών τροπολογιών. Ευχαριστώ το σημειώνουμε. Συμβαστική α υπέρ. Όχι, με συγχωρείτε. Προφορική τροπολογία. ECR. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική α χωρίς την προφορική. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική β, β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 95 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 96 υπέρ κατά τα αποχές απερίφθη 97 υπέρ κατά και επαληθεύουμε την 97 Πέρασε. Εγκρίνεται 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 100 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε. Μάλλον έχει εγκριθεί. Πέρας. Εγκρίνεται 101 υπέρ. Κα, υπέρ. Κατά. Άποχες. Επαληθεύουμε. Βλέπω κάποιες ανάμεικτες τοποθετήσεις από τις ομάδες, με προηγούμενες. Άρχισε πληροφορία λοιπόν. Πέρας και εγκρινεται 2,15 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική ή ε υπερκατα κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική F σίγματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται GZ υπέρ κατά αποχές 156 υπέρ κατά αποχές και απερίφθη 163 υπέρ κατά αποχές απερίφθη H τα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 561 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επαληθεύουμε 561 πέρας εγκρίνεται συμβαστική I, θ δηλαδή, υπερκατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική J, Ι, υπερκατά αποχές εγκρίνεται, 193 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε αρχίζει η ψηφοφορία Πέρασε. εγκρίνεται συμβαστική για το α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 200 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Παρακαλώ να σας βοηθώ να έρθει. Με συγχωρείτε για την διακοπή. Συμβαστική M, τα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. N, δέλτα υπέρ κατά γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο, δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Π, ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Q, τα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 307 υπέρ κατά και επαληθεύουμε 307 πέρας και εγκρίνεται Συμβαστική T υπερκατά αποχές εγκρίνεται. U υπερκατά αποχές εγκρίνεται. V με προφορική τροπολογία υπερκατά, αποχές. Τι θέλατε. Θέλω να εξηγήσω την προφορική τροπολογία. Εξ να εξηγήσετε αφού εγκρίθηκε. Αλλά γράψτε ένα γραμματάκι στους φίλους σας, στους συναδέλφους σας. 362 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 364 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 365 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 370 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 372 υπέρ κατά Αποχές επαληθεύουμε 372 αρχής ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. 374 υπέρ κατά. Αποχές απερίφθη. ΑΑ συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 397 υπέρ κατά αποχές απερίφθη αβ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται AC ε ΑΓ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 399 υπέρ κατά και επαληθεύουμε 399 Vote is closed Τέλος ψηφοφορίας. Α, ισοπαλία, άρα απορρίπτεται. Αλφα δέλτα συμβαστική, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 407 τροπολογία υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 408 υπέρ, κατά. Μάλλον απορρίπτεται, αλλά στο ελέγξουμε καλού κακού. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. 26 υπέρ και 27 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία ΑΕ. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΕΦ. Υπέρ, κατά, αποχέ. Εγκρίνεται. 433 τροπολογία. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ. Απορρίπτεται. 434 υπέρ, κατά, αποχέ. Απορρίπτεται. 435 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 457. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AK υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ΑΛ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 506. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 506 έρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 507. Ποιο είναι υπέρ, κατά, απόχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία α μη, υπέρ, κατά, Κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 522. Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. 559 υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία α μη, υπέρ, ε, α υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 532 υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 532. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και απορρίπτεται. Τροπολογία 535. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία αόμικρον. Ποιος είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 563. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, περνάμε στα έχοντας υπόψη. Ας ψηφίσουμε την 1 έως 4 αρχικό κείμενο από κοινού. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Τροπολογία 1 και 2. 3 και 4 είναι ταυτόσιμες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, Ηλεκτρονικό έλεγχο για τις τέσσερις τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία Εγκρίνονται. Οπότε το αρχικό κατα... κείμενο καταπίπτει. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για το αρχικό κείμενο. Άρχεται η ψηφοφορία. Στο θεωρώντας 7. Δεν ψήφισαν όλοι ακόμα. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται το αρχικό κείμενο στο 7. 27-22. Αρχικό κείμενο το 8. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 10. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο το θεωρώντα 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 με 13 μαζί. Ποιο είναι υπέρ. 10 με 13 θεωρώντας. Κατά αποχές εγκρίνονται. Έχουμε δύο αρχικά κείμενα για το 12 και 13 όχι την τροπολογία 13, το αρχικό κείμενο του θεωρώντας 12 και 13. Εγκρίνονται λοιπόν. Πάμε στην τροπολογία 11. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά αποχέ. Εγκρίνεται. 14 θεωρώντα υπέρ. Κατά. Το άλλο είναι κατά όχι υπέρ. Άρα εγκρίνεται. Τώρα πάμε στην τροπολογία 14. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο του θεωρώντας 15. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και απορρίπτεται 28 ήταν κατά και 25 μόνο υπέρ. Πάμε στο αρχικό κείμενο της 16, του 16 θεωρώντας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 θεωρώντας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο αρχικό κείμενο του θεωρώντας 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 18 υπέρ κατά Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 18 άρχιτη ψηφοφορία. 25 ε, υπέρ, 28 κατά απορρίπτεται. ΑΠ υπέρ εγκρίνεται. AQ ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AR ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εγκρίνεται. Συμβαστική AS υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AT υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, συμβαστική AU υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά Ηλεκτρονικό έλεγχος για την τροπολογία 38. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 24 υπέρ και 21 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικό έλεγχος και για την τροπολογία 39 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ισοψηφία απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία AV. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. AW. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 50. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται. 26 υπέρ, 25 κατά. 54, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 55 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 55, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 26, 27 προς 26. Τροπολογία 56. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 56 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με 26 υπέρ και 25 κατά. Τροπολογία 57. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος και για την 57 άρχεται ψηφοφορία. Ε, πλησιάζουμε προς το τέλος, φαίνεται κάποια κόπος ήδη. Μινοριακές ψηφοφορίες. 27 κατά απορρίπτεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 59. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος απορρίπτεται. Τροπολογία 60. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο του κειμένου όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Και εγκρίνεται με 40 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 7 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή Χωνάς Φερνάντες. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε στο σχέδιο γνωμοδότησης που αφορά τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη-μέλη της άσκησης των εφαρμοστικών εξουσιών της Κομισιόν. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβασμός α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμό 2 υπέρ κατά, τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε επί τη πρόταση όπω αυτή τροποποιήθηκε. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. 49 υπέρ, 4 αποχές και τώρα η δεύτερη γνωμοδότηση για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Διαθεσμικής Συμφωνίας για την καλύτερη νομοθεσία. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές. Να το επαληθεύσουμε παρακαλώ. άρχισε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 με προφορική τροπολογία. Κύριε Λάμπερτ έχετε το λόγο παρακαλώ. Ναι κύριε Πρόεδρε, εμείς είμαστε κατά ε, του να ψηφίσουμε ε, ε, αυτή την προφορική τροπολογία. Ε, αποδυναμώνει τόσο πολύ το κείμενο που πια δεν έχει νόημα. Δεν σημαίνει τίποτα proper transferency. οπότε η ομάδα μας είναι κατά της ψηφοφορίας, ε, κατά, κατά της, της ε, προφορικής ε, τροπολογίας. Εντάξει, θα ψηφίσουμε το συμβασμό 6 χωρίς την προφορική τροπολογία στην περίπτωση αυτή υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε παρακαλώ Πέρας ψηφοφορίας. Εδώ υπάρχει ένας βοηθός που πατάει κουμπιά. Πολύ ενδιαφέρον. Είναι νέα πρακτική αυτή στην Επιτροπή μας. Ε, θα ήταν αρκετά παράνομο ε, Μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένος. Ναι, εδώ, μία βοηθός του ECR, σύμβουλος, άρχισε να πατάει κουμπιά. Συγγνώμη, μπορείτε να πείτε στους ευρωβουλευτές να κάνει το τάδι το δίνα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει στη θέση τους. Mistakes have to be corrected by the MEPs and not by advisors. Chairman, if I may. Ότι λάθο πρέπει να το διορθώνουν οι βουλευτέ και όχι οι βοηθοί. Ε, ο κύριο Σόζα, ξέρετε, δεν μιλάει αγγλικά και θέλαμε να πει γρήγορα η ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή. Ε, δεν υπήρξε κακή πρόθεση. Αν θέλουμε να κάνουμε σκηνέ, υπάρχουν και πιο σοβαροί λόγοι. δεν έχετε το μικρόφωνο. Δεν σας ακούω. Ναι, ως πολιτική ομάδα. Εμεί είμαστε υπέρ τη διαφάνειας προφανώς. Τώρα να κάνετε ολόκληρη σκηνή και κάτι τόσο αστείο, μας ξέρετε νομίζω κάπω καλύτερα. Ήταν πραγματικά ένα λαθό λάθο. Μιλάμε για ένα βουλευτή που δεν μιλάει αγγλικά. Ναι, ο κύριο Χέις και μετά θα πω και εγώ κάτι. Ναι, επί τη διαδικασία Πρόεδρε, το θέμα ήταν το κατώ... αν υπήρχε κατόφλι, κατόφλι, φτάσαμε στο κατόφλι. Τέσσερα άτομα. Για την προφορική τροπολογία, μάλιστα. Ναι, οι τέσσερι πράσινοι. Επιτάχυνα διότι είδα τέσσερα άτομα που ήταν κατά. Ιδάλλως θα κάνει κάτι άλλο. Ε, λοιπόν, θα, να σας πω το εξής. Είναι ατυχές αυτό που συνέβη. Ε, δεν μπορεί οποιοδήποτε άλλος από τα μέλη ε, να πατήσει το κουμπί, έτσι. Το ξέρουμε αυτό, καταλάβαμε βεβαίως γιατί συνέβη, αλλά εφόσον έγινε αυτή τη τελευταία ψηφοφορία, παρακαλώ να επαναληφθεί αυτή η ψηφοφορία για το θέμα αυτό, διότι δεν θέλω ε, να λαμβάνει η χώρα ψηφοφορία ε, με την οποιαδήποτε υποψία ότι κάποιος άλλος ψηφίζει πέρα από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και δεν πρέπει να επαναληφθεί σε καμία περίπτωση. Υπάρχει διερμηνία. Εάν θέλετε, να μου στήσετε ε, να τα πω πιο αργά, θα τα πω πιο αργά. Ε, επίσης, αν υπάρχει πρόβλημα με το κατάλογο, μπορεί η ομάδα να μας το πει για να είμαστε βέβαιοι ότι τα μέλη είναι ενημερωμένα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει όμως και είναι τελώς απαράδεκτο είναι να ψηφίσει κάποιος το όνομα ενό μέλους. Λοιπόν, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 6 χωρί την προφορική τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας Λοιπόν, εγκρίνεται. Συμβασμός Β, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10, με προφορική τροπολογία, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12, υπέρ. Κατά να το επαληθεύσουμε παρακαλώ. Προπολογία 12. Όχι ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε. 13. άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβασμός Γ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά α θα πρέπει να το παληθεύσουμε αυτό 22 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 23 υπέρ κατά να το επαληθεύσουμε το 23 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορία. εγκρίνεται ψηφίσουμε επί του συνόλου τώρα το κείμενο που τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία άρχιτη ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. 47 υπέρ, 0 κατά, 6 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Και τώρα θα περάσουμε στο σχέδιο γνωμοδότησης του Λούντεκ Μαγερ για την ετήσια έκθεση για τις οικονομικές δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Είμαστε έτοιμοι. Πολύ ωραία. Συμβασμός Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός Γ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Με προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. Άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. Υπέρ. Κατά. Να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβασμός Δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός J. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός K. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός L. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 75. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός O υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός P με μια προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ κατά 89. Ε, να το επαληθεύσουμε. Τροπολογία 81. Άρχεται ψηφοφορία. Άρχισε ψηφοφορία είπα, έτσι, ψηφίστε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβιβασμός Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε. Τροπολογία 100 άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 27 ε, κατά 26 υπέρ απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε επί του συνόλου του κειμένου που τροποποιήθηκε με την ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 44 υπέρ, 4 κατά, 5 αποχές. Εγκρίνεται η έκθεση συγχαρητήρια στον εισηγητή. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να κλείσουμε για σήμερα το πρωί θα τα ξαναπούμε ξανά στις 2.30. Στις 2.30 ευχαριστώ.